Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Yeah. Καλό σας απόγευμα. Παρακαλώ καθίστε. Καθυστερήσαμε ήδη πέντε λεπτά. Καλώς ορίζω καταρχήν τους προσκεκλημένους μας. Οι οποίοι θα μας ε, παρουσιάσουν την γνώμη τους τις ιδέες τους, τη γνώση τους σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό για την ε, εργασία του κυρίου Μιλάνα, του αντιπρόεδρου μας, ο οποίος έχει αναλάβει το θέμα της ηχθειοκαλλιέργειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Μιλάνα να κάνει μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, ε, προσκεκλημένους μας. Κύριε Μιλάνα. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Γιατί είμαστε εδώ. Διότι η πολιτική της Ενώσεως τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό απεδείχθη πολιτική που πέτυχε ελάχιστα αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια σε αυτό τον τομέα διαπιστώσαμε μια ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 7 με 8% και ανάπτυξη εντός ενώσεως που δεν ξεπέρασε το 1%. Και γι' αυτό εμείς χαιρετήσαμε θετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζήτησε το Κοινοβούλιο μία τοποθέτηση. Θέση όσον αφορά τη δημιουργία μιας νέας βιώσιμης πολιτικής για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργιών. Περνάμε από αυτή τη λογική, τη βασική λοιπόν, ότι η Ευρώπη τι είναι να δημιουργήσει συνθήκες για να έχει πιο επίκαιρη πολιτική. Πρέπει να κάνει σε αυτό το τομέα πολύ ευαίσθητες επιλογές. Τίποτα δεν αποκλείται σε αυτό το τομέα. Οι επιλογές που θα πρέπει να γίνουν είναι επιλογές ευαίσθητε, διότι αφορούν την αλή από τη μία πλευρά και από την άλλη το περιβάλλον, του καταναλωτέ, την αγορά. Αφορούν πολλού τομεί οι αποφάσει. άρα χρειάζεται στάθμιση προσεκτική των θέσεων για να διαπιστωθεί πόσο, πώς δημιουργούνται οι συνθήκες, οι ρυθμιστικές των κοινοτικών πολιτικών, οι συμπεριφορές των διαφορών κρατών μελών, οι τοποθετήσεις, η στάση του τομέα όλα αυτά να δώσουν θετικά αποτελέσματα. Είναι σημαντική ευκαιρία η σημερινή, διότι καλέσαμε εμπειρογνώμονε που δεν πρέπει να ακούσουν εμένα τόσο που εγώ είμαι ο και τελειώνω αυτό το έγγραφο, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να μα δώσουν και άλλα σημεία προς προβληματισμό. Η θέση μα σήμερα, η θέση μου σήμερα είναι μια θέση ακρόαση περισσότερο, θέλω να ακούσω παρά να δηλώνω πράγματα. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν κάποια σύντομα στοιχεία, αυτό θεωρώ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς η δουλειά που έγινε μέχρι τώρα στην Επιτροπή πέτυχε κάποιους στόχους. Ήδη είπα, μεταξύ άλλων, και η Λισαβόνα και η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο βέβαια διαφορετικό ρόλο εν συγκρίση με το παρελθόν. Η φάση που έχουμε μπροστά μας είναι μια φάση που μπορεί να οδηγήσει σε πρωταγωνιστική θέση το Κοινοβούλιο. Η δουλειά που κάναμε θα πρέπει κανονικά να δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποιες κατευθύνσεις. Γύρω από δύο, τρία, τρία τέσσερα μάλλον βασικά θέματα. Μιλάμε για καλλιέργεια. Μιλάμε για τρόφιμα, για παραγωγή τροφίμων που συνδέεται με την αλληλεία και είναι άμεσο αποτέλεσμα των θαλασσίων δραστηριοτήτων, αλλά μην υποτιμούμε ότι αυτό γίνεται και σε γλυκό νερό. Και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες των ειδών που έχουμε τα ψάρια, έχουμε τα διάφορα όστρακα, έχουμε τα ψάρια του γλυκού νερού, οπότε έχουμε διάφορα είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις. είναι πάντα μικρότερε οι πηγές, οι πόροι της παραδοσιακή αλίας. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περισσότερο. Τα αποθέματα, τα αλλιευτικά στη θάλασσα αποτελούν αντικείμενο όλο και περισσότερων ρυθμίσεων. Γιατί, διότι το δυναμικό εν συγκρίση με την αυξανόμενη ζήτηση για την κατανάλωση ψαριών στον κόσμο ε, αντιμετωπίζουν κίνδυνο οι πόροι, τα αποθέματα. Και κάτι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε, ότι η κατανάλωση των ψαριών είναι 5.500 τόνοι το χρόνο των ψαριών του γλυκού νερού και η εξωτερική κατανάλωση δεν ξεπερνά 1.200.000 τόνοι. Δηλαδή ούτε το 20% δεν καλύπτει η παραγωγή της ε, ζήτησης. Οπότε πώς συνδέεται με την μηχανισμοί, πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της αλληλευτικής πολιτικής αυτά είναι κεφαλαιόδους σημασίας θέματα για τη δουλειά που κάνουμε. Μεταξύ άλλων, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μια μορφή αμοιβαίας μεταφοράς εργατικού δυναμικού από κάποιες δραστηριότητε που αλλιευτικές παραδοσιακές, το εργατικό δυναμικό από βιομηχανική αλλιευτική δραστηριότητα, εργατικό δυναμικό που μπορεί να μεταφερθεί από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Οπότε, η ένταξη της υδατοκαλλιέργειας εντό τη πολιτική που ακολουθούμε για την αλληλεία είναι κάτι που είναι σημαντικό σαν επιλογή. Μετά, ποια είναι η σχέση με του καταναλωτέ. Σημαντικό θέμα. Όσον αφορά αυτό το θέμα, έχουμε ένα στόχο να ανακτήσουμε ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή παραγωγή. Υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση σήμερα και τόσο μεγάλη κατανάλωση στην Ευρώπη και εσωτερική παραγωγή τόσο χαμηλή. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικού λόγου. Πρώτο λόγο είναι ότι υπάρχει επιθετικότητα των εισαγωγικών των διεθνών αγορών έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, που αυτή η επιθετικότητα οδηγεί σε εύκολη εισαγωγή. Γιατί το λέω αυτό. Η ανταγωνιστικότητα των εξ των προϊόντων των εκτός Ευρώπης είναι πολύ υψηλότερη. Τώρα δεν θα αναφερθώ στι λεπτομέρειε. Όλοι καταλαβαίνετε του λόγου για του οποίου ε, που κρύβονται πίσω από αυτό. Κόστο παραγωγή, έλλειψη ελέγχων, ε, υγειονομικέ συνθήκε υπό τι οποίε μεγαλώνουν τα ψάρια που διαφορετικά τα δικά μα. Υπάρχει μια σειρά λόγων. Εμεί θα πρέπει να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Λοιπόν, οδηγό των εργασιών μα είναι η ποιότητα. Η ποιότητα του Ευρωπαίου παραγωγού, του Ευρωπαίου ε, προϊόντος είναι ένας μοχλός μέσω του οποίου μπορούμε να ανακτήσουμε και την ανταγωνιστικότητα. Και μετά και ρύθμιση των εισαγωγών. Άλλο θέμα. Αλλά πιστεύουμε ότι η στρατηγική της Ενώσης θα πρέπει να είναι μια στρατηγική η οποία τίνει να δώσει ποιότητα, να προωθήσει την ποιότητα του ευρωπαϊκού προϊόντος για να δώσει στο προϊόν αυτό μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει αυτή η αντίληψη, αυτή η εικόνα, αυτή η ιδέα να είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης θετικής των καταναλωτών και να δημιουργηθούν πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση που να επιτρέπουν να απολύεται αυτό του είδους η εικόνα, η ποιοτική. Αυτή η εικόνα περνά μέσα από πράγματα που σημειώνται στα τρόφιμα, από στοιχεία, ανιχνευσιμότητα του προϊόντος. Ένα από τα στοιχεία ε, που δημιουργούν εμπιστοσύνη για το προϊόν η δημιουργία πολιτικής σημάτων ή βιομηχανικών προϊόντων, αλλά πάνω απ' όλα των βιολογικών προϊόντων. Και αυτό είναι μια επιλογή προϊόντων ποιότητα, προέλευση. Ή δράσεις ανάντι που είναι δράσεις της τομεακής οικονομίας που αυξάνουν όμως την ανταγωνιστικότητα και την αντίληψη του καταναλωτού. Δηλαδή να βλέπει ο καταναλωτής ότι βρίσκεται ενώπιον ενώπιον ενό προϊόντο που μπορεί να είναι πιο ακριβό, αλλά έχει εγγενή ε, αξία μεγαλύτερη από τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν, αν είναι σαφείς οι κανόνες, εάν έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική, αν τα ακολουθήσουμε αυτά θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες έναντι των εισαγωμένων προϊόντων. Σήμερα είναι άνισες οι σχέσεις, εντελώς άνιση σχέση προσφοράς και ζήτησης. Οπότε τα προϊόντα το προϊόν εισαγωγή είναι στο τραπέζι μα χωρί να υπάρχουν τα αναγκαία χέγγια, ούτε να υπάρχει ε, να ασκούνται αναγκαία έλεγχοι. Δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό που αναφέρθηκε στι εφημερίδε. Ε, είχαμε το, τα προϊόντα τα βιετναμικά. Κανεί δεν ξέρει τη μορφή του προϊόντος που φτάνει. Αν πρέπει να ρωτήσουμε εκτό από του εμπειρογνώμονε, ρωτήσαμε πώ arriva già bello sfilettato. Λοιπόν, πώς έρχεται αυτό το ψάρι εδώ, τι μορφή, το αντιλαμβάνετε το παγκάσιο σαν ένα τρόφιμο, σαν να είναι παράγωγο του προϊόντος ε, τη της αλίας. Δεν ξέρω, ένα είδος τσιμπούρας. Είμαι περίεργος εγώ προσωπικά πώς είναι αυτό το ψάρι το Βιεταμέζικο που μοιάζει με τσιμπούρα Και όμως ε, κατέκτησε την οτροπία της. Α, το ξέρεις. Α, ο αντιπρόεδρο Στίβενσον θα μας πει ακριβώς, θα μας κάνει μια περιγραφή λοιπόν λεπτομερή αυτού του ψαριού. Πρέπει να πω ότι το προϊόν κατέκτησε ε, σημαντικά μέρη της αγορα. και ξεσκεφτείτε ότι είναι, είναι προϊόν του ποταμού Μεκόγκ. που δεν ξέρουμε καν ε, τι γίνεται, τι ρίχνονται, ε, τι μέτρα καθαρισμού του ύδατος του ποταμού κόγκ ε, υπάρχουν. Και αν καθαρίζει το νερό. Υπάρχει και τρίτο θέμα σημαντικό που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργιών έχουν συνέπειες όσον αφορά το περιβάλλον, το γύρο περιβάλλον. Σημαντικό αντίχτυπο. Υπάρχει πρόβλημα συμβίωσης με την τουριστική δραστηριότητα και άλλες δραστηριότητες οικονομικές. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχέσεις με το περιβάλλον το γύρο λόγω καταλήπων, ε, λόγω τροφίμων που διαχέονται. Υπάρχει φυσικός αντίκτυπος αλλά και αόρατος αντίκτυπος που επηρεάζει το περιβάλλον. Ποια είναι η ιδέα που διαμορφωθήκε στο μυαλό μου ότι πρέπει να μιλάμε για ένα ρυθμιστικό, γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις θάλασσες ή ποιε δυσκολίε ανάπτυξη σχετίζονται με την ευκολία με την οποία μια εγκατάσταση υδατοκαλλιέργεια μπορεί να ενεργοποιηθεί. Όλα αυτά απορρέουν από περίπλοκες νομοθεσίες, από έλλειψη εναρμόνισης και απορρέουν αυτά και από μια αρνητική αντίληψη. Κάθε φορά βλέπει κανείς κάποια υδατοκαλλιέργεια δημιουργεί μια εικόνα για το αν θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να ανοίξει σε συγκεκριμένο μέρος. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να ανοίξει το δρόμο. Μέσα από αυτό το δρόμο θα πρέπει να καθοριστούν ακριβείς αυστηροί κανόνες, προϋποθέσεις. Δηλαδή ότι η θάλασσα μπορεί να, να αντιμετωπιστεί σαν κάτι μπορεί να σχεδιαστεί. Όπως και στις πόλεις. Έχουμε... Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρομοίως και τη θάλασσα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τις αναγκαίες συνθήκες για το σχεδιασμό εκμετάλλευσης της θάλασσας. Να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Τι καλλιέργεια έχουμε υπόψη μας. Μπορούμε να έχουμε ιδετοκαλλιέργεια η οποία να, ε, να είναι κοντά στην ακτή όπου μικρής κλίμακας. Να έχουμε πολλές μικρομεσές επιχειρήσεις που έχουν μικρό αντίκτυπο. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας κάνει έρευνα για offshore εγκαταστάσεις, υπεράκτιες, με τη χρήση αιωλικών μορφών ενέργειας, ε, να υπάρχουν μεγάλες εξωτερικές πλατφόρμες για υδατοκαλλιέργειες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες λοιπόν και συσχετισμοί. Η υδατοκαλλιέργεια, παράκτια, βιομηχανική, υπεράκτια, ε, μικρής κλίμακας, μεγάλης κλίμακας, παράκτια, υπεράκτια κλπ. για να μειωθούν οι συνέπειες. Και κάτι αλληλένδετο είναι και η διατροφή και η υγεία των ζώων. Επ' αυτού θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Α, ακριβώς, διότι γύρω από το πρόβλημα, το προηγούμενο, η, η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι και αποτέλεσμα του πώς μεγάλωσε το ψάρι, πώς ζουν τα ψάρια ουσιαστικά στην υδατοκαλλιέργεια. Άρα είναι και θέμα πυκνότητας ύδατος, ζώων στο, νερό, πόσα είναι, και θέμα διατροφής είναι η παλιά ιστορία. Θα το αναφέρω στα γρήγορα λοιπόν. Το, το, το μεγάλο ψάρι το, το μικρό, το ένα ψάρι το, το άλλο. Άρα υπάρχει μια φιλοσοφία που λέει για να μεγαλώσουμε ένα χιλιόγραμμο υδατοκαλλιεργίας χρησιμοποιούμε 2 κιλά ή 3 κιλά ψαριών για διατροφή αυτών των ψαριών, πιθανότατα δεν κάνουμε καλή δουλειά ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τη θάλασσα, ούτε για τους καταναλωτές. Αυτή η ιδέα λοιπόν θα πρέπει να απορριφθεί. Δεν αντιμετωπίζω τις συνθήκες εδώ. Πρώτα απ' όλα, διότι πόροι, που προέρχονται από τη θάλασσα χρησιμοποιούνται διαφορετικά. Το έχω πει στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την ιδέα να χρησιμοποιούμε άλευρα, ηχθιά άλευρα ή ηχθιέλαια για να μεγαλώνουν αγελάδες. Να τρέφονται αγελάδες. Και μετά να μην έχουμε αλευρα για να μεγαλώσουμε τα ψάρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα συνολικό διασύνδεσης μηχανισμών και της όλης οικονομίας, αλλά το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Το αναφέρω διότι δεν υπάρχουν μόνο μία μορφή απόψεις. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Εγώ αναφέρω κάποιες σκέψεις για να ανοίξουμε κάποια διαδρομή, κάποια πορεία στη σκέψη μας και να τα έχουμε υπόψη. Λοιπόν, κλείνοντας, ποιος είναι ο στόχος της δουλειάς που κάνουμε θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε κατεύθυνση όσον αφορά τι στρατηγικέ που συνδέονται με το περιβάλλον, με του καταναλωτέ, με την αλληλεία, με την ανανέωση, την αναζωγόνηση τη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να τα κάνουμε αυτά λαμβάνοντα υπόψη δύο στοιχεία βασικά. Το πρώτο στοιχείο. Προσπάθεια να δημιουργήσουμε κανονισμό για την ιδετοκαλλιέργεια ενιαίο που θα συμπεριλαμβάνει τις δεκάδες επί δεκάδων προδιαγραφές, τις εκατοντάδες προδιαγραφές που σήμερα βρίσκονται σε διάφορους κανονισμούς. Κάποιοι από αυτούς αφορούν τη γεωργία. Ε, σκεφτείτε ότι η βιολογική δατοκαλλιέργεια έχει έναν κανονισμό στον οποίο παραπέμπει. Κανονισμό που αναφέρεται στη γεωργία, όπου έγινε προσωμείωση της ε, διατροφής των ψαριών και της, ε, των καλλιεργιών των βιολογικών. Και όλο αυτό το πλαίσιο ξεκινά από την προπόθεση ότι ο βιολογικό τομέα, όπω θα μα πούνε και οι δικοί, είναι ένα τομέα όπου θα πρέπει να προωθήσουμε αυτόν τον τομέα, να δημιουργήσουμε προοπτικέ. Οπότε σχετική νομοθεσία με τη βιολογική διδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Θα πρέπει να πούμε στον κανονισμό που είναι ενήμερος είναι καινούριο, καθορίζει στόχου, αλλά εμπεριέχει όλα αυτά που ακολουθήθηκαν για την υδατοκαλλιέργεια ψηρά ετών στην Ευρώπη. Ο δεύτερο πυλώνα όσον αφορά την νομοθεσία είναι να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο, συγκεκριμένο ταμείο. Εδώ στην υδατοκαλλιέργεια δαπανώνται πολλά χρήματα. Δαπανώνται όμω από την έρευνα, από τη γεωργία, από άλλου τομεί τα παίρνουμε. Να υπάρχει ένα ενίο ταμείο ειδικό ταμείο ενδεχομένω ή ένα ταμείο εντός του, του, του μέσου για την αλληλεία αλλά να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και να μπορεί να συνδράμει στην επίθεση των στόχων. Και αν υπάρχει ένα λόγος για τους οποίου τα τελευταία χρόνια οι άλλοι αναπτύχθηκαν και εμείς μείναμε ε, στο ίδιο σημείο είναι για, ίσως για αυτό το λόγο. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έτσι συνολικά, να βρούμε μια απάντηση μέσω πολιτικών με τους κατάλληλους πόρους. Επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Εγώ ήδη μίλησα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιλάνα. Θα δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, Φερνάντο Οτέρο Λαουρίδο, διευθυντής της Αρόγα. Είναι μια ένωση παραγωγών καλκανιού στη Γαλλικία. Κύριε Οτέρο Λαουρίδο, έχετε το λόγο. Καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λόγια του κύριου Μιλάνα ε, εμπνέουν άμεσες απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, ε, θέλω να ακολουθήσω λίγο τη σειρά την οποία είχαμε προβλέψει. Συνεπώ θα, θα σας κάνω την παρουσίασή μου και μετά, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σχολιάσω και αυτά τα οποία έθιξε ο κύριος Μιλάνα. Δεν, σε, δεν φαίνεται πολύ καλά αυτή η διαφάνεια, αλλά θα έπρεπε ε, να, είναι, ε, να έχει χρώμα κόκκινο αυτή η διαφάνεια. Ε, έντονο χρώμα. Γιατί όταν μιλάμε για καλλιέργεια στην Ευρώπη, είμαστε σίγουροι όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Ο κύριος ε, Μιλάνα μίλησε για τη ε, διαδικασία διαμόρφωσης καινούργια νομοθεσία τομέα και τα, που, που συμπίπτει χρονικά με ένα μεγάλο αριθμό κρίσιμων σημείων, έτσι τα ονομάζω εγώ, που πιέζουν και συμπιέζουν τον τομέα. Στην ε, Ευρώπη ως ευρωπαϊκή χθιοκαλλιέργεια μπορούμε να θεωρήσουμε δύο πράγματα. Δηλαδή έχουμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Ή θα δεσμευτούμε να αναπτύξουμε μια αποδοτική κερδοφόρα και ευρωπαϊκή χθιοκαλλιέργεια ή δεύτερη εναλλακτική λύση ε, η σταδιακή εξαφάνιση του τομέα στην Ευρώπη υπέρ τρίτων εξοκοινωτικών χωρών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκινώντας από την ανακοίνωση τη ε, επιτροπή προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ε, βλέπω ότι έχουμε δύο, ε, τέσσερις, τέσσερα σημεία σημαντικά. Πρώτον, βιωσιμότητα, που χωρίζεται σε ποιότητα υδάτων, επιλογή των τόπου των εγκαταστάσεων και η προστασία των αρχών της φύσης. Δεύτερον, δεύτερος άξονας της ανακοίνωσης, στήριξη και αποδοχή όλων. Τρίτον, το level playing field, δηλαδή οι, οι ισότιμοι κανόνες συμμετοχής. Και τέταρτον, η υγεία των ζώων. Για αυτά τα τέσσερα θέματα έχω να πω το εξή. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, να σας ε, δώσω το παράδειγμα, θα σας δώσω το παράδειγμα της Γαλλικίας, σε εξηγήσω τι κάνουμε εκεί σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα της θεοκαλλιέργειας. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε καταφέρει και θα συνεχίσω με ελπίζω να το καταφέρνουμε, να διατηρούμε και τις ε, τρεις αυτές διαστάσεις της βιωσιμότητας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο άξονα, υποστήριξη και αποδοχή όλων, νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι σωστή, με όλο το σεβασμό μου. Αν ξεκινούμε, ξεκινήσουμε τη βάση ότι η ηχθειοκαλλιέργεια πρέπει να αρέσει σε όλους, Τελείω η ηχθειοκαλλιέργεια. Πάντοτε θα υπάρχει κάποια ομάδα οικολόγων, όχι όλοι, κάποιοι, και κάποια ομάδα γειτόνων, και πάλι όχι όλοι, που σίγουρα θα διαφωνήσουν. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε στην Ισπανία και ιδιαίτερα στη Γαλλικία με ομό τρόπο. Υπάρχουν κάποιες μειοψηφικές ομάδες οι μειοψηφούσες ομάδες που ε, αντιτίθενται πολύ έντονα στην ανάπτυξη τομέα και πράγματι την παραλύουν. Σε ό,τι αφορά την τρίτη ανησυχία, το τρίτο ζήτημα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ισότιμη συμμετοχή, ε, έλεγχο των εισαγωγών με βάση συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις παρόμοιες με τις προϋποθέσεις που έχουμε εμείς η παραγωγοί στην Ευρώπη, συμφωνούμε πλήρως, είναι ένα σημείο κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση το οικονομικό κλειδί της βιωσιμότητα του τομέα. Σε ό,τι διαφορά το, την υγεία των ζώων, συμφωνώ. Υπό την περιπτώση ότι θα γίνει μια προηγούμενη τεχνική ανάλυση για να αποφύγουμε προκαταλήψεις και μαξιμαλιστικές, πολλές φορές ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις που συχνά δεν ταυτίζονται με την λογική της πραγματικότητας. Το έγγραφο λοιπόν μιλάει ε, για την συνέργεια, την ποιότητα των ε, υδάτων και την ε, βιωσιμότητα. Το ερώτημά μου είναι, είναι δικαιολογημένες αυτές οι ανησυχίες. Να σας δώσω το παράδειγμα της Γαλλικίας. Στην Γαλλία ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Ε, εμείς εκτός από τα μύδια έχουμε ως δεύτερο βασικό προϊόν το καλκάνι. Έτσι, για αυτά τα δύο είδη μιλάμε κυρίως. Ε, προσπαθούμε να σεβαστούμε πάρα πολύ αυστηρά ε, τις αρχές το, της φύσης, ιδιαίτερα το Nature Web και ε, διενεργούμε αυστηρούς ελέγχους σε ό,τι αφορά τα απόβλητα προκειμένου να διατηρήσουμε την ποιότητα των υδάτων. Όπως σας είπα, έχουμε ένα σύστημα ε, εγκαταστάσεων στο έδαφος, χερσαίων εγκαταστάσεων. Όπως σας είπα, ε, εδώ και καιρό ασκούμε μια πολύ προγραμματισμένη ε, ηχθειοκαλλιέργεια. Εδώ και 8-10 χρόνια έχουμε ξεκινήσει. Αυτός ο προγραμματισμός, ο χωροταξικός προγραμματισμός γίνεται σε τομεακό επίπεδο, κλαδικό επίπεδο στο σύνολο δηλαδή του κλάδου. Ε, θεωρούμε δηλαδή τον κλάδο ενοποιημένο, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις πτυχές του, όλους τους, ε, όλους τους κλάδους. Και αυτό το χωροταξικό σχέδιο ε, καθορίζει πού μπορεί να γίνει θεοκαλλιέργεια, με ποιο τρόπο και σε ποιο μέγεθος. Μέσω ενός νόμου που είναι ένα χωροταξικό σχέδιο κατά βάση. Είναι ο νόμος που προβλέπει το χωροταξικό σχέδιο. Ο στόχο, η στόχη αυτού του σχεδίου είναι να επιλεγούν οι κατάλληλες από τεχνικής πλευράς ζώνες για την ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας ε, στο έδαφος και δεύτερον ο καθορισμός των γενικών αρχών που θα διέπουν αυτή την ηχθειοκαλλιέργεια των ε, κανόνων. Εμείς συγκεντρώσαμε σε συγκεκριμένα πολύγωνα αιθιοκαλλιέργεια στη αν θέλετε, τα μέρη στα οποία είναι δυνατόν να επιτραπεί η ηχθειοκαλλιέργεια στη στεριά. Συγκεκριμένες ζώνες λοιπόν, συγκεκριμένα πάρκα ή πολύγωνα. Και δεύτερον, δεδομένου ότι το χωροταξικό προβλέπει στο συγκεκριμένο σημείο ε, την εγκατάσταση ε, ηχθειοκαλλιεριών, ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται δηλαδή η εγκατάσταση ε, ε, ηχθειοκαλλιέργειας σε, σε όλα τα υπόλοιπα εδάφη. έτσι ώστε οι ηχθειοκαλλιέργειες να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες ζώνες. Επίσης, ε, καθορίζουμε τους κανόνες τους οποίους λειτουργούν και δημιουργούνται οι ηχθειοκαλλιέργειες και τρίτον, ε, πώς είναι δυνατόν να προστατεύσουμε το περιβάλλον ε, εξασφαλίζοντας την τριπλή ε, βιωσιμότητα του περιβάλλοντος βέβαια, την κοινωνική και την οικονομική. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια περιοχή απομακρυσμένη από το κέντρο και ακόμα και οι περιοχές της είναι απομακρυσμένες σε σχέση με το κέντρο της Γαλλικής δεν έχουν πολλέ ε, υποδομέ, ενδεχομένω οι υποδομέ του είναι οι υποδομέ που κατασκευάζονται για τι ηχθειοκαλλιεργίε. Έχουμε καθορίσει δύο τύπου κριτηρίων. Τεχνικά κριτήρια και ε, πολεοδομικά κριτήρια. Με βάση αυτά γίνεται μια συγκεκριμένη επιλογή επί των προτάσεων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Ορισμένες από αυτές γίνονται δεκτές, άλλες από αυτές απορρίπτονται. Έτσι έχουμε πράξει ως τώρα. Λοιπόν, καταρχήν μίλησα για τεχνικά κριτήρια. Είναι προφανές ότι για να εξασφαλίσουμε την θεοκαλλιέργεια καλκανιού στο, στη στεριά. Ε, η θερμοκρασία παράδειγμα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 20 βαθμούς ε, ή να πέφτει κάτω από τους 10 ω 12. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις. Ε, υψόμετρο, περιεκτικότητα σε άλλα κλπ. Το πρόγραμμα αυτό είναι συμβατό με το δίκτυο Natura, αλλά ε, το αποφεύγουμε. Έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε τις ε, εγκαταστάσεις αυτές μέσα σε ζώνες του δικτύου Natura. Ε, Παρ' όλα αυτά λέω ότι το σχέδιο αυτό είναι συμβατό εκτός και αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προστασία της συγκεκριμένη ζώνης. Μετά, έχουμε τα πολεοδομικά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή διακρίνουμε μεταξύ δύο, τύπου εγκαταστάσεις, δύο τύπων εγκαταστάσεις. Αυτές που είναι ε, επεκτάσεις παλαιότερων και τις νεότερες εγκαταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις, με βάση αυτό το ε, σχέδιο, στη Γαλλικία μπορούν να κατ' εξαίρεση να γίνουν επεκτάσεις σε περιπτώσεις προστατευμένων ζωνών αλλά ποτέ σε, σε ζώνες που υπάρχουν οικοσυστήματα προτεραιότητας. Οι νέε εγκαταστάσει όμω δεν μπορούν να γίνουν σε καμία ζώνη προστατευόμενη, ούτε καν σε προστατευόμενε ζώνε. Ούτε στο δίκτυο Natura, ούτε πουθενά. Συνοψίζοντα λοιπόν, στην Γαλλική υπάρχουν 24 πάρκα ή πολύγωνα ακτιοκαλλιέργεια. Έχουν προβλεφθεί με σύμφωνα με το ισχύον προσχέδιο 11 επεκτάσει και 13 καινούριε εγκαταστάσει, Στο δίκτυο Natura 3 επεκτάσει, παλαιότερων εγκαταστάσεων, καμία νέα εγκατάσταση, ενώ βέβαια σε οικοσυστήματα προτεραιότητα καμία απολύτω εγκατάσταση. Τώρα, το σχέδιο αυτό κάνει διάκριση μεταξύ εγκαταστάσεων ε, σε κανονικής προστασίας σε εγκαταστάσεις σε κανονικής προστασίας ζώνες και ε, εγκαταστάσεις σε μέγιστης ή αυξημένης προστασίας ε, ζώνες σε κανονική προστασία ζώνε ε, η, η κάλυψη μπορεί να είναι τα 2 τρίτα, μέχρι τα 2 τρίτα του συνολικού εμβαδού. Ε, και επιτρέπονται δύο όροφοι με συνολικό ύψος 7 μέτρων. Ε, σε περίπτωση ζωνών αυξημένης προστασίας, ειδικής προστασίας, προβλέπεται ένας όροφος και 3,5 μέτρα ύψος. Όπως σας είπα είχαμε κριτήρια αποδοχής και κριτήρια απόρριψης με βάση τα οποία γίνεται δεκτή μια πρόταση ή απορρίπτεται μια πρόταση. Έχουμε τέσσερα, τέσσερις ομάδες κριτηρίων. Περιβαλλοντικά, ε, πολεοδομικά, βιολογικά και κοινωνικά. Καταρχήν λέμε ποια είναι τα κριτήρια απόρριψης, με βάση τα οποία γίνεται απόρριψη. Δηλαδή, ε, αμέσως και αυτόματα ε, απορρίπτεται μια πρόταση ε, όταν ε, προβλέπεται εγκατάσταση χθιοκαλλιέργειας σε περιοχές με αμολόφους, σε περιοχή του, περιοχές του δικτύου Natura με οικοσυστήματα προτεραιότητας ή εκεί που είναι μοναδικό το περιβάλλον. από πλευράς πολεοδομικής δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις σε ζώνες αστικές ε, ή που έχουν προβλεφθεί να ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως. Το βιολογικά κριτήρια ε, ε, Έχουμε, δεν πρέπει να είναι κοντά σε ζώνες ε, που έχουν ε, αυξημένη μόλυνση Και, λοιπά. και κοινωνικά κριτήρια να μην είναι κοντά σε τουριστικές ζώνες, ε, να μην ενοχλούν αισθητικά, οπτικά κλπ. Εδώ πέρα βλέπετε την πρώτη θαλάσσια, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο προστασίας στη Γαλλικία. Είναι το, σημείο το οποίο θεωρήθηκε ε, βέλτιστο ως προς την ποιότητα των υδάτων, τους, των υδάτων του. Πριν από έξι χρόνια το ζήτησαν ήδη ίδιοι Είναι ε, πάρκο προστασίας των θαλασσίων ειδών. Λοιπόν, εδώ και 20 χρόνια συμβιώνει αυτή η περιοχή με μία από τις μεγαλύτερη, στην τρίτη μεγαλύτερη εγκατάσταση ηχθειοκαλλιέργειας στη Γαλλικία. Ε, εδώ και 18 χρόνια βρίσκεται αυτή η εγκατάσταση. Ε, αντλεί, χρησιμοποιεί και απορρίπτει νερό, 3 κυβικά μέτρα κατά 3 ε, κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο για 18 χρόνια. Και παρόλα αυτά συμβιώνει αυτή η εγκατάσταση με το θαλάσσιο πάρκο ε, αριστερά εδώ βλέπετε ότι είναι το χωριό βλέπετε πάνω την εγκατάσταση και τις, ε, τις ε, ξόδους του νερού ε, απόρριψης του, των υδάτων της εγκατάστασης δεξιά. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα των αποβλήτων. Εδώ και 20 χρόνια το κάνουμε. Αυτή είναι η ίδια εγκατάσταση. Βλέπετε ότι δεν προσβάλλει οπτικά αισθητικά. Βλέπετε ότι το ύψος των κτηρίων συμπίπτει με το ύψος, με το υψόμετρο του, της γης γύρω. Δηλαδή βλέπετε την κόκκινη γραμμή από την ε, από το δρόμο ή από την ε, γη δεν φαίνεται η εγκατάσταση αυτή γιατί έχουμε σκάψει στο έδαφος, έχουμε χτίσει οπότε το ύψος το οποίο φτάνει το κτίριο, φτάνει τα κτίρια δεν ξεπερνάει το ύψος του δρόμου. Αυτό μπορεί να γίνει. Έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται στη Γαλλικία. Αυτό όμως υπό την προπόθεση ότι όλες οι δυτικές υπηρεσίες συνεργάζονται και έχουν μια αποφασιστικότητα, μια πολιτική βούληση να αναπτυχθεί η χθιοκαλλιέργεια. Αναρωτιέται κανένας γιατί έχουμε τόσα κρίσιμα σημεία, τόσες κρίσιμες πλευρές στον τομέα μας. Δεδομένου ότι ο χρόνο μα πιέζει να πω ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι η άγνοια. Άγνοια από πλευρά του πληθυσμού, από πλευράς ορισμένων πολιτικών και από ορισμένων υποτομέων που σχετίζονται με τη θάλασσα. Ταυτόχρονα ε, κάποιοι ε, χρησιμοποιούν με, για δικό τους όφελος της, ε, την πληροφόρηση την χειραγωγούν συγκεκριμένα, τη μανιπουλάρουν. Τρίτον, υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ε, κυβέρνηση ή προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται μακρινή, θεωρείται κάτι καινούριο και θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετό βάρος στην γεωστρατηγικο-οικονομική ισορροπία. Σε ό,τι αφορά το κράτος ή τις περιοχές του, τις περιφέρειες του, οι ε, πολλοί πολιτικοί τοπικοί θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν δυσάρεστοι στο κοινό τους, στους πιοφόρους τους. Παρόλο ότι ε, γενικά οι διαφωνούντες είναι λίγοι, παρόλο ότι κάνουν πολύ θόρυβο. Ταυτόχρονα και ε, οι πολιτικοί αλλά και οι διοικητικές αρχές πολύ συχνά ε, θεωρητικά υποστηρίζουν την ε, οχθιοκαλλιέργεια. Κανένας δεν έχει πει ποτέ, δεν έχω ακούσει εγώ ποτέ, κάποιον να λέει ε, δεν πρέπει να αναπτυχθεί η οχθιοκαλλιέργεια. Όχι, δυστυχώς όμως, στην πράξη αυτές οι γενικόλογες δηλώσεις δεν ακολουθούνται από συγκεκριμένες πράξεις, κίνητρα και αποφασιστικότητα. Υπάρχει βούληση αλλά δεν υπάρχει αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα για να επιτύχουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να σώσουμε την ηθιοκαλλιέργεια για το μέλλον. Δεύτερον, να τη δώσουμε επαρκή χώρο να αναπτυχθεί. Δηλαδή, ε, μετά, διαδικασίες ε, ασφαλείς, ταχείες, αποτελεσματικές και ασφαλεί. Και τρίτον, ένα σύστημα που θα επιτρέπει τον έλεγχο των εισαγωγών, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται με τα ίδια κριτήρια και με τις ίδιες ευκαιρίες που γίνεται η, η κοινωτική παραγωγή. Γιατί ευρωπαϊκή ηχθειοκαλλιέργεια. Ε, είναι στερεότυπο αυτό. Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αγορά σε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα για το ψάρι. Ε, σιγά σιγά αυξάνουμε όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε πιο μεγάλες ποσότητες από αυτές που παράγουμε εμείς. Και βέβαια η Ευρώπη είναι ένας χώρος πολύ έντονης επιστημονικής προσπάθειας. Εμείς έχουμε ένα Ινστιτούτο και είμαστε οι πρώτοι που ε, επιτύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι πρώτοι λέω, για ένα εμβόλιο εναντίον παρασίτου τα ψάρια. Μια τέτοιου είδους επιτυχία απαιτεί σημαντική προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης. Ε, δεν θέλουμε αυτή η ανάπτυξη να γίνει εκτός των ευρωπαϊκών, η έρευνα και ανάπτυξη να γίνει εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Τι ζητάμε ή ποια είναι η ερώτηση που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Εγώ ξεκινώ από την εξή ε, ερώτηση. Θέλει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί η, η δατοκαλλιέργεια. Γιατί εδώ και πολύ καιρό αναπτυσσόμαστε πολύ αργά, αργά, αργά και, όλο και, πιο, και με όλο και πιο πολλά προβλήματα. Αν πούμε ότι δεν θέλουμε ε, την ηχθειοκαλλιέργεια, εντάξει, εκεί τελειώνει η συζήτηση, σιγά σιγά θα κλείσουν οι εγκαταστάσεις, ε, θα μειωθεί ο αριθμός τους μέχρι να μηδενιστούν. Εμείς έχουμε ήδη μια τραπεζική εγγύηση προκειμένου να, να επαναφέρουμε το τοπίο στην αρχική του κατάσταση αν κλείσουμε. Γίνεται αυτό. Ε, η ηχθειοκαλλιέργεια θα γίνεται σε τρίτες χώρες. Εκεί θα αναπτυχθεί σε τρίτες χώρες και από τρίτες χώρες και μετά εμείς θα εισάγουμε ψάρια για μάλιστα ε, εκτός των δικών μας παραδόσεων. Το σχολείο ο κ. Μιλάνα. Ε, το θέμα το, του, του Βιετνάμ και του κατά πόσον καθαρίζονται τα νερά του Μεκόγκ. Δεν γίνεται να καθαρίσουν τα νερά του Μεκόγκ. Γιατί το νερό αυτό δεν κινείται. Παίρνουν μια τεράστια ποσότητα νερού. Ε, το τοποθετούν σε ένα πηγάδι. Εκεί μεγαλώνουν τα ψάρια. Και όταν τα ε, πάρουν... Ε, βγάζουν το νερό, ξεραίνεται το νερό, εν πάση περιπτώσει, και τη λάσπη τη χρησιμοποιούν για λίπασμα. Εμεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια πράγματα στην Ευρώπη. Μετά, πολιτική αποφασιστικότητα και υποστήριξη. Ναι, πρέπει, ε, αν θέλουμε την ηχθειοκαλλιέργεια, να διαθέτουμε ένα επαρκές νομικό πλαίσιο, λέω, ε, επαρκές και αποτελεσματικό, ε, που θα επιτρέπει την ε, ηλική και οικονομική ανάπτυξη του τομέα μια ενοποίηση, απλοποίηση ε, της νομοθεσίας με βάση την τριπλή ε, ε ένα, μια αποτελεσματική κοινή οργάνωση των αγορών. Εμείς ε, στην Ισπανία έχουμε μια εξωτερική νομοθεσία για την ε, ε τικετοθεσία, για τη σήμανση. εξαιρετική νομοθεσία. Αυτό που Θέλουμε όμως είναι να εφαρμόζεται και όλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν αποψυχεί, αποκαταψυχθεί και πουλιώνται ως νοπά. Αυτή τη στιγμή η, σήμανση δεν ε, είναι αποτελεσματική. Και τέλος, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανασκέφτεται, αλλά σίγουρα χρειάζεται ε, βελτίωση και διατήρηση των ε, υπαρχόντων ε, υπαρξών εγκαταστάσεων. Μια κοινή οργάνωση αγοράς Πρέπει να τελειώσετε λοιπόν πολύ, έχετε ξεπεράσει την ώρα σας. Ναι, ένα τελευταίο πράγμα. Πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της ε, αμοιβαιότητας ε, ε, στις εισαγωγέ μας και να εφαρμόσουν τα ίδια κριτήρια με αυτά που εφαρμόζουν εσωτερικά. Λυπάμαι, λέει πρόεδρος, ε, πρέπει να σας πιέσω λίγο γιατί έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς χρονικούς. Ο λόγος στον κύριο Μάρκο Γκρέκο, επιστημονικός σύμβουλος της AIAB, Ιταλικής Ένωσης Βιολογικής Γεωργίας. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά για μένα να είμαι εδώ. Για να συμβάλλω και εγώ στη συζήτηση περί βιολογικής γεωργίας. Άκουσα ήδη παρεμβάσεις του κυρίου Μιλάνα και του συγητού που προηγήθησαν και έδωσαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω ένα όραμα να σας παρουσιάσω του βιολογικού που παρουσιάζει, αντιπροσωπεύει την αριστεία το βιολογικό προϊόν. Την αριστεία της βιωσιμότητας στην Ευρώπη ήδη από το 1991. Το βιολογικό προϊόν στην, Ελλάδα, στην Ευρώπη συγγνώμη, σύντομα θα γιορτάσει τα 20 χρόνια του, του χρόνου από πλευράς νομοθετικής. Επιτρέψτε μου εν συντομία να παρουσιάσω την Ιταλική Ένωση Βιολογικής Ιδατοκαλλιέργειας που εκπροσωπώ σήμερα είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με τη βιολογική καλλιέργεια που λειτουργεί από το 1983 και καθορίζει τις προδιαγραφές. Είναι μια ένωση για τον καθορισμό προδιαγραφών και σε υπουργικό επίπεδο. Είναι μια ένωση που έχει περίπου 10.000 μέλη, παραγωγούς, τεχνικούς, καταναλωτές έχει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς του βιολογικού τομέα με άλλα λόγια στους κόλπους της. Έχει ομοσπονδιακή δομή, έχει κεντρικό γραφείο στη Ρώμη, αλλά είναι παρούσα εργάνωσή μας σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας με δομές αυτόνομες σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητε της ενώσεώς μας είναι προθήσεως της βιολογικής γεωργίας έναντι παραγωγών και καταναλωτών. Ενημέρωση κάνουμε όσον αφορά τεχνικές πτυχές ρυθμιστικές πτυχές όσον αφορά την εφαρμογή της μεθόδου της βιολογικής παραγωγής και διάφορες υπηρεσίες που παρέχουμε και κυρίως δραστηριότητε εκπροσώπησης και προστασίας στα διάφορα θεσμικά όργανα, εθνικά και κοινοτικά. Και είναι και μέλος της EFAM, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Κινημάτων της Βιολογικής Γεωργίας. Μεταξύ των δραστηριοτήτων μπορούμε να υπενθυμίσουμε κάποιες εθνικές εκστρατείες, ημερίδες ενημερώσεως των καταναλωτών, όπου εκεί προτείνονται βιολογικά προϊόντα. Κάνουμε να καταλάβουν οι καταναλωτές ποια είναι τα χαρακτηριστικά του βιολογικού προϊόντος που πρόκειται να αγοράσουν και που πρέπει να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά όταν ε, φέρουν το σήμα το κοινοτικό. Κάνουμε και εκδόσεις Ανακοινώσει στον τύπο, στι ιστοσελίδε, ε, έχουμε και εφημερίε ηλεκτρονικέ newsletter και δίνουμε και βραβεία για την ε, βράβευση της αριστεία στην παραγωγή τη Ιταλία. το μέλι, τα κρέατα, το χείριο κρέα κλπ. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που ήθελα να υπογραμμίσω είναι και συμμετοχή των, ε, της Ένωσης σε διάφορα προγράμματα εθνικά σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση του βιολογικού προόντος, η κοινωνική γεωργία. Να υπενθυμίσουμε ότι η βιωσιμότητα είναι και βιωσιμότητα κοινωνική για όλους εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίζουν πρόβλημα μπορεί η γεωργία να παρουσιάσει κάποια ευκαιρία και μετά έχουμε και το τμήμα το περιβαλλοντικό. Δηλαδή θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις, την δύο και τις σχετικές πρωτοβουλίες σε διάφορα εθνικά επίπεδα. Και έχουμε διάφορες δραστηριότητες ερευνητικές στα πλαίσια των προγραμμάτων πλαισίων. Εγώ ανήκω στην Επιστημονική Επιτροπή της Ενώσεώ μας που ασχολείται με την παρακολούθηση της πρόθεσης της έρευνας και τις διάφορες δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης προς τους παραγωγούς, δηλαδή προς, του ε, προς φορεί τοπικούς φορείς και τους τοπικούς παραγωγούς η οργάνωσή μας ε, συνέβαλε στη δημιουργία ενό ιδρύματος, Ιταλικού Ιδρύματος για την έρευνα στην ε, βιολογική γεωργία που λειτουργεί σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο. Ποιε είναι οι εμπειρίες από τη βιολογική παραγωγή και τι σχέση έχει με την ιδετοκαλλιέργεια. Το έλεγε ο κύριος Μιλάνα πριν. Μιλάμε για βιολογικό με τον κανονισμό 710 του 2009, αλλά η Ευρωπαϊκή Δετοκαλλιέργεια υπάρχει από πιο παλιά, από τις αρχές της χιλιετίας. Το 2001 λήξαν τα πρώτα μέτρα, αλλά υπήρχε διάφορα, διάφορες ρυθμίσεις σε κοινοτικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το association και διάφορα άλλα. Υπάρχει ενδιαφέρον σεβασμός του γεωργικού κόσμου που ασχολείται με την βιολογική παραγωγή για να προσεγγίσει επίση με τον ίδιο τρόπο και την υδατοκαλλιέργεια. Όλο το κίνημα που αναπτύσσεται είναι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις και στους διάφορους φορείς και στους διάφορους άξονες, τον τρίτο και τον τέταρτο άξονα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που ήδη έχουν αναφερθεί και υπογραμμιστεί. Άριστα μάλιστα. Και το ανέφεραν και προλαλήσαντες. Σίγουρα χρειάζεται να δοθεί προπτική στο βιολογικό. Με αυτούς που ασχολούνται με τον έλεγχο και την πιστοποίηση της βιωσιμότητας πρέπει να προσεγγίσουν στο θέμα. Και μπορούμε να βεβαιώσουμε και να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχουν εσφαλμένα συστήματα, λαθασμένα συστήματα, τουλάχιστον σε γενικό επίπεδο, αλλά οι τρόποι με τους οποίους τα συστήματα εφαρμόζονται υπάρχουν εκεί τα λάθη. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει βούληση, πολιτική βούληση, κοινοτική βούληση, ε, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για να επιφέρει τις αλλαγές και των κρατών μελών. Να υπάρχει βούληση, λέγω, να πάμε προς βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια βασικά σημεία χωρίς να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες να υπογραμμίσω κάποια πράγματα που ήδη τονίστηκαν. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα έλλειμμα, ένα deficit όσον αφορά τη παραγωγή στην υδατοκαλλιέργεια. Πρόβλημα της μειώσεως της αλληλευτικής προσπαθίας. Της μείωση των διαφόρων πόρων των ηχθείων. Τι μπορούμε να τονίσουμε, τη βιωσιμότητα χρειαζόμαστε. Δηλαδή βιώσιμη αλληλεία και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια χρειάζεται. Και η βιολογική πτυχή που εκπροσωπεί την αριστεία της βιωσιμότητας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου βιώσιμου συστήματος. Αυτό είναι κάτι που ήδη εν υπάρχει στην κοινότητα, στην κοινωτική προσέγγιση. Υπάρχουν διάφορες πτυχές που μπορούν να είναι σημαντικές όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ιδετοκαλλιέργειας. Πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει υπερεθνική, διεθνής πρόθεση που θα συνδέεται αυτή με πολιτικές τομεακές. Είναι σημαντικό λοιπόν η στρατηγική, η πολιτική στρατηγική, η κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί να λαμβάνει υπόψη την προσέγγιση που έγινε σύνθημα λίγο πολύ στον τομέα της υγείας From the farm to the fork, δηλαδή από την καλλιέργεια στο πυρούνι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση. Να υπάρχουν μέτρα υποστήριξη που θα προταθούν, στήριξη τη παραγωγή. Να κάνω μια σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στο βιολογικό τομέα. Χρηματοδοτούνται οι επιχειρησει οι εκμεταλλεύσει εκεινε αυτε δημιουργούνται και αναπτύσσονται και χρηματοδοτείται ε, η χρηματοδότησή του προωθήσει 10 χρόνια μετά τη δημιουργία του. Και γινόταν αυτό 10 χρόνια μετά τη δημιουργία όταν δεν υπήρχαν πλέον ε, εκμεταλλεύσει. Χρειάζονται λοιπόν τα κατάλληλα μέτρα και οριζόντια και κάθετα. Ολοκληρωμένα μέτρα, συντονισμένα μέτρα για να βοηθούν τι επιχειρήσει. Η ενημέρωση του καταναλωτού είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Πρέπει ο καταναλωτή να ξέρει να έχει εμπιστοσύνη στο προϊόν τη βιώσιμη ιδετοκαλλιέργειας. Σε αυτό θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και μέτρα υποστήριξης, μέτρα πολιτικής στήριξης και οικονομικής στήριξης των διαφόρων τομέων. Αν θέλουμε βιώσιμη δατοκαλλιέργεια, βιολογική καλλιέργεια. Η ανταγωνιστικότητα υπενθυμίστηκε από τον Ισπανό συνάδελφο προηγουμένως Πιστεύουμε ότι περνάει ανταγωνιστικότητα μέσω τη αξιοποίησεω τη ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια, τη αξιοποίησεω των αυτοχθόνων ειδών. ήδη που έχουν αξία, εγενή αξία, που συνδέεται με τη διατήρηση της βιοπικιλότητας και τη διατήρηση των τεχνικών διατροφής, αλίευσης, που έχουν συνέπειες οικονομικές και κοινωνικές όλα αυτά, επιτόπιες όσον αφορά τα παραδοσιακά αυτά είδη που αλλιεύονται. Υπάρχουν ελλείψεις που ήδη υπογραμμίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Καλλιέργεια, καλλιεργεία κυρίως, ζωοτεχνικές πτυχές έχουν και ένα, δηλαδή αναπαραγωγή, ανατροφή, διατροφή μάλλον. Και η διατροφή των ζώων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη βιωσιμότητα, την οικονομική των υδατοκαλλιεργειών. Αυτό σίγουρα είναι κάτι επί το οποίο πρέπει να βασιστούμε και προς τα εκεί να ερευνήσουμε διεξόδους. Άλλο θέμα, θέλουμε έρευνα που να έχει αντίκτυπο όχι βραχυπρόθεσμο, με βράχη μέσο πρόθεσμο, με προγράμματα τα οποία να συνδέονται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας επιτόπου, δηλαδή καινοτομία και μεταφορά γνώσης που είναι άλλη πολύ σημαντική πτυχή. Ο τομέας της αλληλεία, της θεατοκαλλιέργεια, ε, είναι ένα τομέα πολύ προχωρημένος που κάπου όμως έχει κενά σε κάποιες περιοχές. Μπορεί η έρευνα να βοηθήσει να στηρίξει τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Άλλη σημαντική πτυχή είναι της αξιοποίησεως της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας. Και εδώ έχουμε την εμπειρία της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Αξιοποιούμε τι σημαίνει, να εντοπίσουμε, να γνωστοποιήσουμε ένα προϊόν. Δηλαδή, τομεακή προσέγγιση. Το προϊόν, τι κατεύθυνση θα ακολουθήσει στην αγορά, τι προορισμό. Η αξιοποίηση μπορεί να περάσει μέσω του ορισμού ενός σήματος που παρέχει εχέγγυα. Βάσει κριτηρίων θα δίνεται αυτό το σήμα. Ελάχιστα κριτήρια θα μπορούσαμε να πούμε διότι είναι ένας τομέας περιπλοκότατος, πολυπίκυλος, οπότε υπάρχουν πολλά είδη, πάνω από 350 είδη που διατρέφονται, πολλά είδη παραγωγής. Χρειάζεται ένα σήμα με ελάχιστα κριτήρια στα οποία θα βασίζεται. Όσον αφορά την γεωργία, την βιολογική υπάρχει ήδη αυτό, διότι η γεωργία ήδη έχει ενσωματώσει, το είπαμε, όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, έχει συμμορφωθεί μέσα σε ένα κανονισμό. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα. Αυτή την περίοδο υπάρχει διάδοση διαφόρων σημάτων, υπάρχουν πολλά είδη πιστοποίησης που απευθύνονται στην ίδια, ή παρόμοιες μεθόδους παραγωγής και στην ίδια αγορά. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια έναντι του καταναλωτού. Θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα κριτήρια, κυρίως ελάχιστα κριτήρια περιβαλλοντικού χαρακτήρα και θα πρέπει να έχουμε και οικολογικό σήμα, όπως το Eco Label, οικολογικό σήμα, που μπορεί να προωθεί αυτό το σήμα την αναγνωρισιμότητα και των προϊόντων της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, αλλά και, τις, και τα προϊόντα της βιώσιμης αλίες Εντός ποιου πλαισίου μπορούμε να κινηθούμε για να εντοπίσουμε τα ελάχιστα κριτήρια. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση, νομοθεσία, όπως στον τομέα της επιστημιστικής ασφάλειας, την ασφάλεια των τροφίμων. Πέρασε η περίοδος των οδηγιών και ο κανονισμός τώρα είναι το απλούστερο, το πιο εύκολο μέσο που αμέσως εφαρμόζεται τα κράτη-μέλη. Η δατοκαλλιέργεια είναι ένα τομέα περίπλοκος, πράγματι. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε όλες τις ιδιαιτερότητες εθνικές και τοπικές ιδιαιτερότητες. Χρειάζονται όμως ελάχιστα κοινά κριτήρια που θα φορούν όλα τα κράτη-μέλη για να πιστοποιούν το προϊόν και να υπάρχει ισοδυναμία σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Κάποια κριτήρια θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμού τοπικού. Αυτό αναφέρθηκε ήδη για τη Γαλλικία. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, εάν δεν κάνω λάθος. Χωρικού σχεδιασμού Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αφορούν την Ιταλία. Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό των διαφόρων τόπων εσωτερικής υδατοκαλλιέργειας. Σχέδια χωροταξίας, όπως η Λιγουρία και η Σικελία. Να εντοπίζεται λοιπόν προδιαγραφές χωροταξίας που θα οδηγούν σε μια ε, κοινωνική βιώσιμη προσέγγιση να μπορεί να συμμετέχει η περιοχή, να συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι stakeholders, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο και θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνεπειών, του αντικτύπου. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να εντάσσονται σε ευρύτερο κριτήριο ολοκληρωμένης διαχείρισης της υπαίθρου της περιοχής. Θα μπορούσε να αποκληθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να αξιολογηθούν κάποιε φυσικέ περιοχέ περιθωριοποιημένε, αλλά κυρίω ούτω ώστε να υπάρχει διάδραση θετική σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ υδατοκαλλιέργεια και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, παραδείγματο χάρη τουρισμό, γεωργία. Και με την αλληλεία να υπάρχει επαφή. Η αλληλευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να ενταχθεί. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, διάφορα προγράμματα σε κοινοτικό επίπεδο με δραστηριότητε υδατοκαλλιέργεια σε περίοδο παύση άλλων καλλιεργιών. Αυτά όλα μπορούν να ληφθούν υπόψη και θα ήθελα να σταθώ να πω μερικά ε, λίγα λόγια για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει στην Ευρώπη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και σε αυτή τη φάση ποια είναι η σχέση βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια με βιολογική υδατοκαλλιέργεια. παραθέτω μία ένδειξη που δίνει ο ΦΑΟ που λέει ότι η βιολογική παραγωγή έναντι της πράσινης παραγωγής, της οικολογικής παραγωγής είναι ορισμοί περιορισμένοι που αναφέρονται σε ξεχωριστές πτυχές μεμονωμένες στις βιωσιμότητες. Η βιολογική παραγωγή και η ετικέτα σημαίνει ότι υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής και μεταποίησεως τομεακή προσέγγιση που μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία μέσω διαφόρων προδιαγραφών που θα πρέπει να ακολουθούνται. Είναι ένα σύστημα αριστείας, ένα σύστημα το οποίο δεν θέλει να καλύψει απαραίτητα όλη την κοινοτική υδατοκαλλιέργεια. Μπορεί να έχαμε και ένα πιο γενικό σύστημα κοινοτική υδατοκαλλιέργειας και να μιλάμε για ποιοτική υδατοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από τη μία πλευρά να έχουμε την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και από την άλλη να έχουμε την βιολογική, πιο γενική. Λοιπόν, η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια θα ήταν προαπαιτούμενο της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που ήδη υπάρχει στη γεωργία. Παραδείγματο χάρη μεταξύ ολοκληρωμένη καλλιέργεια, ε, γεωργία και βιολογική καλλιέργεια. Μπορούν να πάρουμε αυτά τα παραδείγματα και όσον αφορά τι σχέσει μεταξύ των δύο προσεγγίσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα, των δύο γραμμών βιωσιμότητα. Και υπάρχουν διάφορε ιδιαίτερε πτυχέ, κάποιε ήδη υπενθυμίστηκαν, που αφορούν αυτέ οι προσεγγίσει, οι γραμμέ, πτυχέ που μπορούν να αξιοποιήσουν την υδατοκαλλιέργεια. Το να μιλάμε για την ε, των ζώων είναι πάρα πολύ δύσκολο, την καλή κατάσταση, την καλή διαβίωση των ζώων. Ε, Προηγουμένω έγινε λόγο για αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε ένα κριτήριο μεταξύ άλλων Δηλαδή η αλληλεία για την αξιολόγηση των προϊόντων. Είναι περίπλοκο τομέα αυτό τη ευζοία των ζώων. Είναι ένα τομέα που δεν υπάρχουν επαρκεί γνώσει ακόμα για να εντοπίσουμε ε, ποια πρέπει να είναι η πυκνότητα διαφόρων τέτοιων ε, εκμεταλλεύσεων. Πόσα ζώα εμπεριέχουν. Θα πρέπει όμω να υπάρχουν τα αναγκαία εχέγγυα για να, υπάρχει, να διατηρείται η ισορροπία του οικοσυστήματο. Να υπάρχουν προσανατολισμοί, κατευθυντήρε γραμμέ που προανέφερα. Ε, το ελάχιστο βάθο, παραδείγματο χάρη, για τι υπεράκτιε καλλιέργειε ή ετοκαλλιέργειε. Ποια πρέπει να είναι η ελέγχου των περιοχών εκείνων όπου ε, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών. Θα πρέπει να υπάρχει ανάντι έλεγχος που προηγείται τις εγκαταστάσεις των υδάτων πριν την εγκατάσταση και ε, ένας έλεγχος του γίνεται το νερό μετά την εκμετάλλευση. Είναι ευαίσθητα όλα αυτά. Άρα πρέπει να έχουμε τη μέγιστη πυκνότητα βάσει ε, διαφόρων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που δεν θα πρέπει να ξεπερνάμε αυτά τα όρια. Ποιες πυκνότητες χρησιμοποιούνται κανονικά στην εντατική υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να δούμε. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν κτηνιατρικά φάρμακα, να χρησιμοποιούνται και διάφορα ειδικά μόρια για την ε, ε, απολύμανση των εγκαταστάσεων και βέβαια και η πτυχή των τροφίμων που χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, η έρευνα πρέπει να γίνει εκεί. Να μειωθεί η ζωική πρωτεΐνη στα τρόφιμα για τα ψάρια στο ΦΑΟ. Αναφέρω ότι περίπου 25% των αλλιευμάτων τελικά είναι διατροφή άλλων ψαριών. Οπότε πρέπει να δούμε τι σχέσει υπάρχουν μεταξύ βιώσιμη ιδετοκαλλιέργεια και βιώσιμη αλληλεία. Διότι από τη βιώσιμη αλληλεία μεγάλο ποσοστό ε, παράγει τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για την ε, διατροφή των ε, ψαριών στι ιδετοκαλλιέργειε. Για να κλείσω. Διότι μου ήρθε και σημειωματάκι σχετικό. Μου λέει να τελειώνω. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, από την εμπειρία του βιολογικού τομέα θα κλείσω λέγοντα τα εξή. Φέτο είδαμε το ότι μπήκε σε κοινοτικό κανονισμό η ε, βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή, ε, πέρασε ας πούμε επισημοποιήθηκε και ε, ορμάνε όλοι πάνω στον τομέα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Θέλουμε ποιοτική υδατοκαλλιέργεια, θέλουμε βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Θα πρέπει η ρύθμιση να είναι αυστηρή θα πρέπει να εντοπίζει περισσότερο, λιγότερες παραμέτρους, αλλά παραμέτρους που θα είναι αυστηρές παράμετροι επιστημονικά και τεχνικά, ούτως ώστε να υπάρχει αξιοπιστία αναφέρθηκε η εικόνα της ποιότητας, η αντίληψη για την ποιότητα. Καμιά φορά ο κατανοτής αντιλαμβάνεται διαφορετική ποιότητα από αυτή που είναι η πραγματική ποιότητα του προϊόντος. Είναι η, αυτή που αντιλαμβάνεται, η αντιληπτή ποιότητα. Θα πρέπει η αντιληπτή ποιότητα λοιπόν να αντιστοιχεί στο ε, στην αριστεία του κοινοτικού προϊόντος. Λοιπόν, θα μπορώ να συνοψίσω τα διάφορα μέτρα που θα έπρεπε να μπουν σε μια νομοθεσία, δηλαδή της αξιοπιστίας αυτό, να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τον κύριο Λεωνίδα Παπαχαρίση, Διευθυντής Ποιότητας ε, της, ε, του Ομίλου Νηρέας. που κυρίως ασχολείται με τσιπούρες αλλά και με άλλα είδη Μεσογείου. 15 λεπτά παρακαλώ. Μέχρι τώρα οι προηγούμενοι προλήσεις δεν σεβάστηκαν το χρόνο. Τους έχετε το λόγο κύριε Παπαχαρίση. Good afternoon, Καλώς απόγευμα. Για να καταλάβουμε την ισχύ της ε, προτυποποίησης. υπάρχει και ένας Έλληνα, μετά τον κύριο Γκρέκο υπάρχει και ένας Γκρέκο Έλληνας που έχει και πιστοποιητικό το διαβατήριο. Σας ευχαριστώ πάρα που μας δώσατε την ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψή μας για το μέλλον του τομέα μας. Δεν θα περιγράψω την ανάπτυξη του τομέα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, μια και οι περισσότεροι από εσά τη γνωρίζετε. Άλλωστε, περιλαμβάνεται και στα έγγραφα εργασία τη σημερινή συνεδρίασης. Να σας ε, μιλήσω για δύο λόγια, με την δική μα εταιρεία. Εμείς παράγουμε το 18% ε, της ε, παραγωγής λαβρακιού και τσίπουρας της Ελλάδας. 19% της συνολικής παραγωγής Μεσογείου. Σήμερα έχουμε μια εμπειρία την οποία θα θέλουμε να μοιραστούμε σε αυτό το επίπεδο το πολυεπίπεδο, πολυεθνικό επίπεδο ε, που ε, σίγουρα θα μας ε, θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια καινούργια νομοθεσία που θα επιτρέψει έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποτελεσματικό αποδοτικό τομέα εχθειοκαλλιέργειας η χθιοκαλλιέργεια ήταν τμήμα της ε, κοινή ε, πολιτικής αλίας πριν από 30 χρόνια ε, αλλά αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να εργαστούμε προκειμένου τα, όχι τα κέρδη μας, τα έσοδά μας τα, ε, τα, τα ωφέλη μάλλον προκύπτουν να ε, συντηρηθούν και στο μέλλον. Δύο χρόνια πριν μόλις προέκυψαν τα πρώτα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν τις αρχές ε, της ε, βιολογικής χθιοκαλλιέργειας, παραγωγής θεοκαλλιεργίας και την υγεία των θαλάσσιων οργανισμών. Εμείς έχουμε κανόνες επίσης και στην καθημερινή μας ε, λειτουργία. Ε, και βέβαια θα πρέπει να λυθούν υπόψη και οι ειδικέ ε, συνθήκε που επικρατούν στο περιβάλλον, οι ειδικέ ιδιότητε των διαφόρων ειδών κλπ. Πιστεύουμε ότι απαιτείται μια ευρωπαϊκή νομοθεσία πλαίσιο για να μειώσουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, της λειτουργίας, την εχνηλασιμότητα και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε την παραγωγή μας έναντι ε, εισαγωγών από τρίτε χώρες που λαμβάνουν χώρα με διαφορετικούς όρους. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίδιους όρους ε, και στα προηγούμενα θέματα που ανέφερα, αλλά και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων, ε, τις, ε, τους κανόνες πεδί ζωοτροφών, την ευημερία των ζώων και την διαχείριση του περιβάλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις, ο τομέας της θεοκαλλιέργειας απουσιάζει από προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές και περιοχές όπου πολλές φορές ε, ε, χαρακτηρίζονται από ένταση σε άλλες δραστηριότητες όπως τουρισμό, αλληλεία κλπ. Ε, η, η, αλήθεια είναι ότι η χθιοκαλλιέργεια δεν χρειάζεται πολύ μεγάλες εκτάσεις και αυτό που χρειάζεται όμως είναι καλής ποιότητας νερό. Και οι άλλες δραστηριότητες θα πρέπει ε, συμπεριλαμβανομένης και της ε, οικοδομής θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ε, η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα μπορεί να εξασφαλίσει ποιότητα των υδάτων, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις διαφορετικές δραστηριότητες εκείνων των περιοχών, στην υποπόσταση ενός μιλίου στην αναθεώρησή της θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, guidelines για την ε, ποιότητα των ε, υδάτων της ηχθειοκαλλιέργειας. Αν η ηχθειοκαλλιέργεια ενταχθεί στα προγράμματα περιφερειακή ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών σίγουρα θα είναι καλό και κοινωνικά ε, για τι παράκτητε κοινότητε. Η υγεία των ζώων ε, έχει αναγνωριστεί πρόσφατα ω ε, μεγάλη σημασία ζήτημα. σε πολλέ περιπτώσει φαίνεται ότι το ζητά η ίδια η αγορά και ενθαρρύνεται από περιβαλλοντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλου ενδιαφερόμενου. Η υγεία των θαλάσσιων ζώων είναι επίση προτεραιότητα οποιασδήποτε χθιοκαλλιεργία. Τα υγιή ζώα αναπτύσσονται πιο γρήγορα, πιο πολύ, επιβιώνουν περισσότερο και βέβαια έχουν καλύτερη σάρκα. Ε, οποιαδήποτε όμως ε, ρύθμιση, νομική ρύθμιση υιοθετηθεί θα πρέπει να ε, ε, υιοθετηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να αποφευθούν σημαντικά εμπόδια, μη επιστημονικά εμπόδια στην ανάπτυξη τομέα. Σε κάθε περίπτωση ε, παρόμοιες απαιτήσει ε, θα πρέπει να επιβληθούν και σε προϊόντα τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Τέλος, αυτές οι πρακτικές, αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και σε άλλους ε, τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική ηχθειοκαλλιεργίας θα πρέπει να υποστηριχτεί οικονομικά, να χρηματοδοτηθεί. Στον κανονισμό τον οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο κονδύλιο για την χρηματοδότηση έρευνας, ε, υιοθέτησης καινοτομίας και ε, επαγγελματικού προσ... επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους ε, ενδιαφερόμενους. Επίσης, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε, σε διαρθρωτικό έργο ε, για να ε, υπηρετήσουν και τα συμφέροντα της ηθιοκαλλιέργειας. Περισσότερες, ε, περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ε, μπουν στον τομέα σύντομα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται καινοτομία και πρέπει να υποστηριχθούν, ε, να δοθεί έτσι μια δεύτερη όθηση στον τομέα της χθιοκαλλιέργειας. Οι, προτεραιότητες, οι ερευνητικές ε, θα πρέπει να εντοπιστούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτές, ιδιαίτερα αυτές που ε, εστιάζονται στην αύξηση του προϊόντος του τομέα. Για παράδειγμα, καλλιέργεια καινούριων ειδών χαμηλές, στα χαμηλά επίπεδα της αλυσίδας, πρωτογενής, δευτερογενής παραγωγή δηλαδή. Αυτό θα αποσυνδέσει το μέλλον της ηχθειοκαλλιέργειας από, τις, ε, από τα, τη, την αλίευση ε, ελεύθερων ειδών από την ε, ανοιχτή θάλασσα. Δεύτερον, πρωτοβουλίες για να υποστηριχθεί η προαγωγή ευρωπαϊκών ειδών σε τόπιο περιβάλλον και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών. Έρευνα για ε, ε, που ε, γίνεται σε μολυσμένα περιβάλλοντα επίσης θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος, θα πρέπει να δούμε και την ηχθειοκαλλιέργεια άλλων ειδών. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ηγέτιδα δύναμη στον επιστημονικό τομέα. Ο βασικός ε, στόχος όμως θα πρέπει να είναι να διαθέτουμε βάσιμα επιστημονικά στοιχεία προκειμένου να, ε, να, να λάβει η χώρα μια εφαρμοσμένη έρευνα. Η Ευρωπαϊκή ε, Ο Ευρωπαϊκός τομέας θα πρέπει να έχει ένα σαφή ρόλο με προτάσεις και προτεραιότητες προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη τομέα. Η πρωτοβουλία για τον ε, καθορισμό ενώ μιας καινούργιας ε, νομοθεσίας πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ηχθειοκαλλιέργεια ε, είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Το κείμενο αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη που θα οθήσει τον τομέα. Δεν χρειάζονται άλλα εξοδικητικά έγγραφα που σχετίζονται με χαμηλότερης σημασίας καθημερινές λειτουργίες και δραστηριότητες. Η Ευρώπη ε, πρέπει να γίνει ένα σημαντικός παίκτη στον κλάδο αυτό, να αναπτύξει τις δυνατότητες και το δυναμικό ε, σε, και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για να το, να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε επιστημονική γνώση υψηλής ποιότητας, τεχνικούς και, έμπειρου ε, και έμπειρους τεχνικούς και επιστήμονες και βέβαια υγιείς επιχειρήσεις που θα είναι ικανές να αναλάβουν τους επενδυτικούς κινδύνους που είναι απαραίτητοι για ένα τέτοιο σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαχαρίση και ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε και το χρονοδιάγραμμά σας. Δύο ακόμη είναι στον κατάλογο, ένας από αυτούς είμαι εγώ. Αλλά θα δώσω πρώτο το λόγο στον κύριο Βαλέσα. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα. Αυτή είναι η ε, λέξη που χαρακτηρίζει την ηχθειοκαλερή, ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη μας στη Λατινική Αμερική ή την Ασία. Καταρχήν όμως θα πρέπει να υποστηρίξουμε επιστημονικά και οικονομικά την χιοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα στην παραδοσιακή χιοκαλλιέργεια που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε είναι η κατάλληλη παρακολούθηση. των ευρωπαϊκών και των εισαγόμενων προϊόντων έτσι ώστε να ακολουθούνται και να επιβάλλονται οι ίδιοι κανόνες. Ακούσαμε από τους ομιλητές κάποια λόγια, αλλά όταν μιλάμε για την διδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Γιατί είναι απολύτως ζωτική ε, σημασία για τον τομέα της υδατοκαλλιέργεια. Μία από τις αρχές της ε, οδηγία αυτή είναι ο σεβασμός και η προστασία των ε, πόρων. Και οι χρήστες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο το νερό που χρησιμοποιεί η υδατοκαλλιέργεια επιστρέφει στο περιβάλλον, δεν καταναλώνεται. Υπάρχουν άλλοι χρήστε που καταναλώνουν το είδο που χρησιμοποιούν. Έχει, α, έχουν ακουστεί προτάσεις για επιβολή τέλους επί του ύδατος που χρησιμοποιείται από την υδατοκαλλιέργεια. Νομίζω ότι εδώ επικρατεί μια παρεξήγηση. Είναι σαν να λέμε ότι θα επιβάλλουμε τέλος για τη χρήση του ατμοσφαιρικού αέρα. Η λίστα πρέπει να αναζητηθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πρόβλημα σωστό. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία είπαν, εισήγαγαν τέλη, ένα ειδικό φόρο, ο οποίος οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ουγγαρία. Λοιπόν, χρειάζονται αρχές σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων, των φυσικών πόρων από την υδατοκαλλιέργεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλέσα. Έγιναν διάφορα σχόλια για την υγεία. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη να τα λάβουμε υπόψη το τομέα της καλλιέργεια. Όπως είπε ο κ. Μιλάνα όμως, το πρόβλημα είναι πως ότι εισάγουμε τεράστιες ποσότητες ψαριών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βαλέσα είπε θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και να εφαρμόζουμε τα ίδια ίδιες προδιαγραφές και τους ίδιους κανόνες. Αλλά οι προδιαγραφές υγείας των ζώων δεν αναγνωρίζονται από τον WTO, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ε, ως επαρκής ε, αιτιολογία για να μπλοκάρουμε κάποιες εισαγωγέ. Συνεπώς, η υγεία των ζώων δεν περιλαμβάνει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Λυπούμε βέβαια, γιατί αν πηγαίνατε στο Δέλτα του Μεκόν και βλέπατε πώς εκτρέφονται τα παγκάσιους, θα διαπιστώνατε ότι οι προδιαγραφές ε, ε, υγεία των ζώων δεν πλησιάζουν καν τις δικές μας. Συνεπώ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτέ. Ίσως το παγκάσιο για αυτούς ε, είναι εξαιρετικά φτηνό ψάρι, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν ε, πως υπάρχει ένα τίμημα που πληρώνουν. Αυτό που ήθελα όμω να σχολιάσω είναι το εξή. Προς τον κύριο Μιλάνα κυρίω. Το θέμα της κλασικής εξίσωσης. Πολλοί λένε ότι ταΐζουμε ψάρια στα ψάρια και ταΐζουμε υπερβολικό ε, χθιάλευρο στα ψάρια και θα πρέπει να εισάγουμε καλύτερα λαχανικά ή ε, κάποιες φυτικές ύλες. Γιατί το σημερινό σύστημα οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των αλληλευτικών αποθυμάτων. Όταν μπήκα σε αυτήν την επιτροπή πριν από 10 χρόνια, ε, το ποσοστό ήταν 70% ηχθιάλευρα και 30% ε, φυτικά άλευρα. Οι επιστήμονες εργάστηκαν και τα ηχθιάλευρα έχουν πέσει στο 40% με 60% δημητριακά. Νομίζω ότι η πρόοδος είναι εξαιρετική. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουμε ψάρια φυτοφάγα. Τα ψάρια τρώνε ψάρια. Δεν είναι δυνατόν η δίαιτά τους να αποτελείται κατά 100% από αλεύρι σόγιας. Το 40-60 νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτή τη στιγμή. Επίσης, πολλοί λένε ότι χρειάζονται 4, 5, ίσως και 6 κιλά ψαριού για να παράγουμε ένα κιλό ε, ψαριού σε υδατοκαλλιέργεια. Δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους τομείς, αλλά στον, τομέα του Σολομού, στη Σκοτία, αυτή τη στιγμή ε, η αναλογία έχει πέσει σε 1,1 κιλό τροφής ψαριού για παραγωγή ενός κιλού ψαριού. Στο, στα πουλερικά η αναλογία είναι 2,5 κιλά προς ένα. 2,5 κιλά ζωοτροφής για ένα κιλό κοτόπουλου. Στον τομέα του, βαϊού, του βοηού κρέατος είναι 7 προς ένα η αναλογία. Οπότε η, ο τομέας υδατοκαλλιέργειας κάνει πολύ καλή δουλειά. Και ας είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας. Αυτά τα λέω για να συζητηθούν. Ίσως αργότερα θα μπορούσα να κάνω κάποια σχόλια για την χρήση των ε, αποβλήτων ε, για, ως τροφή στα, για τα ψάρια. Ευχαριστώ. Το ουσιώδες εδώ για, την, ε, για το μέλλον και για την αύξηση της υδατοκαλλιεργίας είναι αυτή η εξίσωση της, των τροφών για τα ψάρια και τα άγρια είδη ψαριών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ε, ηχθειοτροφών. Όντως δεν υπάρχουν ακόμη φυτοφάγα ψάρια, δυστυχώς. Τα ψάρια όμως όπως ο γάδος, ο σολομός και άλλα ο ερυθρός τόνος που τα καλλιεργούμε σε κλωβούς είναι αυτά που προτιμούμε και εμείς να τρώμε περισσότερο στην Ευρώπη. Ίσως λοιπόν η τεχνολογία να μπόρεσε να βελτιώσει τα πράγματα σε σχέση με 10 χρόνια πριν με, σε ό,τι αφορά την μίξη των λαχανικών σε, στις αλλά ξέρω ότι έχουμε και έναν εκπρόσωπο από την Ορβηγία εδώ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την βιομηχανία του Σολομού και ξέρω ότι ο νορβηγικός Σολομός και η συγκεκριμένη ε, βιομηχανία έχει ε, μια, έχει μια ένα προς ένα στην, ε, στα τρόφιμα, στα, στις τυχθιοτροφές. Εμείς εδώ στην Ευρώπη κάναμε μια έρευνα και ε, είδαμε ότι ο ρυθμός, ε, η σύγκριση αυτή δεν είναι τελικά ένα προς ένα, ακόμη και στην ε, Νορβηγία είναι δύο προς ένα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο όριο του πόσο μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε για την του καλλιέργεια. Οπότε και αυτό είναι σχετικά ανησυχητικό για την βιομηχανία των άγριων ψαριών. Πρέπει να αφήσουμε τα αποθέματα να αυξηθούν ώστε μακροπρόθεσμα να μπορούμε να αυξήσουμε τα αλλιεύματα. Αλλά βραχυπρόθεσμα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτά σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Στίβενσον. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τους εκπροσώπους για τις σκέψεις τους για οικονομικές ενισχύσεις και τις ανάγκες που έχετε εσείς ως προς αυτό. Θεωρείτε ότι χρειάζεστε οικονομική στήριξη για, την, ε, για να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί η βιομηχανία. Θεωρείτε ότι οι συνήθεις μηχανισμοί της αγοράς είναι αρκετοί για να ενισχύσουν τον τομέα της ιδιωτικαλλιέργειας. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν διάφορες ε, τοποθεσίες οι οποίες ε, είναι λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλες για το το καλλιέργεια. Η Νορβηγία έχει όλο αυτό το καθαρό νερό, τα φιόρδ, τους ποταμούς που έρχονται από τα βουνά, που καθαρίζουν τους κλοβούς που υπάρχουν Οπότε δεν υπάρχουν, ε, ή τέλο πάντων υπάρχουν ελάχιστα ε, απόβλητα λόγω του καθαρού αυτού νερού και βεβαίως έτσι διευκολύνεται και η ανάπτυξη του ίδιου του ψαριού, του σολομού. Αλλά σε πιο θερμά ύδατα, εκεί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα με ασθένειες κτλ. Είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε την υδατοκαλλιέργεια και ως πού μπορούμε να την επεκτείνουμε, ας πούμε, στην Ισπανία ή στα νότια μέρη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαχαρίσης μήπως θα ήθελα να απαντήσει, γιατί ξέρω ότι πρέπει και να φύγετε. Thank you. Uh, well. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να απαντήσω την πρώτη ερώτηση για την ανάγκη επιδοτήσεων. Κατά την άποψή μας, οι επιδοτήσεις είναι απαραίτητες κάθε φορά που η Ευρώπη θέλει να προωθήσει ένα τομέα. Η αγορά δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Αλλά Αν θέλουμε να διατηρήσουμε ε, ρυθμούς ανάπτυξης όπως αυτούς που είχαμε πριν από 15 έως 20 χρόνια, πρώτον αυτό, και δεύτερον, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον για τομείς που έχουν υψηλό κίνδυνο, υψηλό επενδυτικό κίνδυνο τότε χρειάζονται οι επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την θέση εγκατάστασης, είναι κρίσιμη σημασίας. Ε, τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να επιλεχθούν οι θέσεις των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Στην Μεσόγειο πια έχουμε μια εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Πολλά εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί για να μετρηθεί η επίδραση ε, της ε, θαλάσσιας χιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον της Μεσογείου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μεσογειακή θαλάσσια Αχθιοκαλέρια έχει μέλλον. Υπάρχουν τόποι με ισχυρότατα ρεύματα, ε, μεγάλα βάθη, άνω των 50, 60, 70 μέτρων, όπου ηχθειοκαλλιέργειες μπορούν να εγκατασταθούν με ασφάλεια και να λειτουργούν χωρίς σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μία μικρή παρένθεση. Για τα παράσιτα, ας πούμε. Αυτό που χρειάζεται για να δημιουργηθούν παράσιτα είναι θερμοκρασία, νερού, νερό και ένα φορέα. Ένα τρίγωνο είναι αυτά τα τρία. Και στι ηχθειοκαλλιέργειες υπάρχουν και τα τρία. Συνεπώς, τα παράσιτα είναι φυσιολογικά στι ηχθειοκαλλιέργειες. Ακόμα άλλωστε και στην ελεύθερη φύση είναι ε, ε υπαρκτά τα παράσιτα. Δεν μπορούμε όμω να πούμε ότι αυτά τα παράσιτα θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία μας. Thank you very much. Indeed, any of the... Ευχαριστούμε. Θέλει κανείς άλλος να απαντήσει? I'm an outsider here, of course. I, we're not in, in the union. Uh, but I, uh, I am a board member of something called... Είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ε, Καινοτομίας και Έρευνας που, στο, στο οποίο συμμετέχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Νορβηγία. Ε, και σίγουρα ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει τον οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε είναι η έρευνα. Δεν είναι δυνατόν να χτίσουμε μια βιώσιμη, ε, ένα βιώσιμο κλάδο ηχθειοκαλλιέργειας χωρίς να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Θα μιλήσω αργότερα για αυτό το ζήτημα. Κύριε Οτέρο Λαουρίδο, Δηλαδή, δύο σχόλια μόνο. Για τις ερωτήσεις της αξιότιμης κυρίας Βουλευτού. Ρωτήσατε, για παράδειγμα στην Ισπανία, πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η θεοκαλλιέργεια. Για τη Γαλλικία μπορώ να σας δώσω το παράδειγμα του τελευταίου χρόνου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο επενδυτικά σχέδια, τα οποία αναμένουν να ε, λάβουν την άδεια ε, μια, ένα, μια καινούργια ευθιοκαλλιέργεια καλκανιού ε, με τρεις ε, υπο ε, 100 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Και μια, ένα άλλο σχέδιο, νορβηγική εταιρεία, που ετοιμάζεται για επένδυση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε ζώνες πάρα πολύ βιώσιμες από κοινωνικής πλευράς. Η καλλιέργεια καλκανιού στο, στη στεριά μπορεί να γίνει ε, σε μια απόσταση τουλάχιστον 3,5 χιλιόμετρων μακριά από οποιαδήποτε αστικό κέντρο. Γιατί ε, υπάρχει πρόβλημα παρασίτων. Τα παράστα βρίσκονται στο νερό. Ε, μπορεί να φτάσουν στη, στη στεριά αλλά δεν δημιουργούνται στη στεριά. Υπάρχουν ήδη από το νερό. Ε, αυτό που είναι πλανκτόν στη θάλασσα γίνεται παράσιτο στη στεριά. Ε, δεν το δημιουργεί το παράσιτο η ίδια η εγκατάσταση. Από την άλλη μεριά, για το θέμα των ε, ζωοτροφών, των τροφών ε, ηχθειοτροφών για την ακρίβεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω τα εξή σχόλια. Ε, ε κάποιες ευρωπαϊκές αρχές ε, θέτουν ως κριτήριο το θέμα των ε, αυτοχθόνων ειδών. Δεν υπάρχουν πολλά αυτοχθόνα είδη που είναι ε, φυτοφάγα. Ελάχιστη στην Ισπανία σχεδόν καθόλου. Δεύτερον, Ε, θα μπορούσε βέβαια να υποκατασταθεί με την έρευνα το κομμάτι των ε, ηχθιαλεύρων που έτσι κι αλλιώς όλο, όλο, και λιγότερο, χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο. Θα μπορούσαμε σταδιακά να αντικαταστήσουμε αυτό το κομμάτι με ε, άλευρα από δημητριακά. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής. Κανένας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που να μπορεί να πιστοποιήσει αυτή την τροφή, άλευρα δηλαδή από δημητριακά, ε, ως μη περιέχουσα ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή ότι ένας παραγωγός ε, ψαριών θα μπορεί να ταΐζει στα ψάρια του άλευρα ε, απαλλαγμένα από γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή ήδη ε, πολλά μεγάλα σούπερ μάρκετ δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή μας διότι φοβούνται ότι στο μέλλον μπορεί να φτάσουν γενετικά τροπημένοι οργανισμοί στην τροφή των ψαριών. Συνεπώς, πώς θα υποκαταστήσουμε τα αλευρά. Οι επιστήμονες εργάζονται επί αυτού. Υπάρχουν όμως και τα ε, ε, ε, συστατικά του αίματος. Ε, ε, μη μυρικαστικών. Μη μυρικαστικών. Ε, υπάρχει ένα ποσοστό, μέγιστο ποσοστό, ε, νομίζω 8%, ε, στο οποίο θα μπορούσαμε να φτάσουμε στις ζωοτροφές. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, κανένας δεν θέλει να, να τα εισάγει αυτά τα παράγωγα αίματος ε, στις ζωοτροφές για λόγους αισθητικού και μόνο. Οπότε πρέπει να γίνει μια επιλογή. Σίγουρα δεν υπάρχει ε, τέλεια λύση. Στην ηχθειοκαλέρια σίγουρα ε, επιβάλλονται πολύ περισσότερε απαιτήσει από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια. Στη Γαλλική έχουμε ένα εκατομμύριο αγελάδε, 400 κιλά κάθε μία. Υπάρχουν όμω μόνο 7 εκατομμύρια τόνοι καλκανιού για πολλούς τα 7 εκατομμύρια τόνοι καλκανιού είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι τα 400 εκατομμύρια τόνοι ε, αγελάδας. Πέραν αυτού βέβαια, ε, τα, οι κριτικές είναι και αβάσιμες, διότι καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι... Καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει ε, κάποια βλαβερή, συγκεκριμένη βλαβερή συνέπεια των ηχθειοκαλλιεργειών στη θάλασσα τόσο των κλοβών όσο και ε, βλάβη που να προέρχεται από την ηχθειοκαλλιέργεια που γίνεται στη στεριά. Εμείς έχουμε ένα αυστηρότατο σύστημα ελέγχου των αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα. Κάθε δύο μήνες ε, κάνουμε, ε, πρέπει να υποβάλουμε έκθεση ποιότητας του νερού, συν τις εκθέσεις που κάνουν και τους ελέγχους που κάνουν οι εθνικές κρατικές αρχές περιοδικά και τακτικά. Συνεπώ, εκπροσωπώ όλε τι επιχειρήσει αυτή τη στιγμή τη Γαλλικία και στην ηχθειοκαλλιέργεια δεν έχουμε ούτε μία καταδίκη ούτε μία καταδίκη, δικαστική καταδίκη για υπέρβαση των ορίων στα απόβλητα. Ενώ για άλλους τομείς έχουμε. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να λέει, να αποδεικνύει ο, με νούμερα, με στοιχεία, ότι τα απόβλητά μας ε, βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Αντιθέτω, υπάρχουν αντίθετα στοιχεία. Συνεχείς αναλυτικές εξετάσεις και αναλύσεις ε, για την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Ε, έχουμε 5 μιλιγράμμ ανά λίτρο. Αυτό είναι το όριο και όλες μας οι αναλύσεις δείχνουν μικρότερα νούμερα στη Γαλλικία, αν βρεθεί μία φορά μία τιμή που να υπερβαίνει το όριο, μπορεί να κλείσουν την εγκατάσταση. Είναι τρομερό ο κίνδυνο. Ποτέ δεν έχει βρεθεί. Μετά, ε, ποιο είναι ο κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί από, υπερβολική, ε, από υπερβολικές αποβλήτων. Ο ευτροφισμός. Δεν το έχουμε δει πουθενά. Αυτό το είδατε η πρώτο, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο προστασία στη Γαλλικία συμβιώνει δίπλα-δίπλα με μία από τις πιο παλιέ εγκαταστάσεις χιοκαλλιέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδατε, είδα ότι φοβάστε μήπω ταΐσετε στα ψάρια γενετικά τροπημένου Οργανισμού. 30 εκατομμύρια όμω τόνοι σόγια γενετικά τροπημένη ε, έχει μπει στην Ευρωπαϊκή, έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ταϊστεί στα ζώα. Το κοινό νομίζει παρόλα αυτά ότι δεν τρώει τίποτα που να έχει σχέση με γενετικά τρομένους οργανισμούς. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα ξυπνήσουμε μία μέρα και θα δούμε ότι οι γενετικά τρομένοι οργανισμοί είναι τμήμα της διατροφής μας, της καθημερινής διατροφής. Ελπίζω να μην είναι πολύ επίμαχο το σχόλιο που έκανα. Ας περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της ε, ακροασής μας θα ήθελα να δώσω το λόγο ξανά στον κύριο Πέτερ Άρνεσεν. Κύριε Άρνεσεν. Mrs. Um, ε, aren't we skipping Mrs. Ε, Dawn Perkins? Δεν ξεχάσαμε την κυρία Dawn Perkins. Sorry. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα και να μπορώ να σας μιλήσω για την καλλιέργεια Σολομού και την εμπειρία της Νορβηγίας. Αυτό μου ζητήθηκε να κάνω, να πω δηλαδή κάτι για το πώς ε, έχουμε δομήσει την δική μας βιομηχανία στην Νορβηγία. Για όσους ξέρουν τη βιομηχανία μας, θα ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε στις, στα τέλη του, της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, αλλά από τις αρχές του 80 η βιομηχανία πραγματικά άρχισε να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς και βλέπετε ότι ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό ταξίδι. Είμαστε ο μεγαλύτερος παραγωγός ε, ε, ε, σολομού στην, στο, στον, στην Ευρώπη, στον κόσμο συγγνώμη, 50% παράγεται στην, στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία ο σολομός είναι το μεγαλύτερο καλλιεργούμενο ζώο. Καλλιεργούμε περίπου 800.000 τόνους σολομού, δηλαδή τρεις φορές της ε, παραγωγής κρέατος, οποιοδήποτε είδους κρέατος. Η παραγωγή έχει, 4 ε, ε, δισεκατομμύρια γεύματα το χρόνο, έχει μια εξαγωγική αξία περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργεί επίσης, επίσης πάρα πολλές θέσεις εργασίας, περίπου 20.000 θέσεις εργασίας συνολικά, αν δούμε και την βιομηχανία παροχής και, στις, ε, και κυρίως ε, για τις ε, περιοχές της Υπέθρου και τις παράκτης περιοχές. Και μάλιστα η τάση είναι να γίνεται η επεξεργασία των ψαριών τοπικά, σε τοπικό επίπεδο περισσότερο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να γίνεται η φιλετοποίηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ μέχρι τώρα έμενε το κεφάλι στο ψάρι, αλλά έβγαιναν τα εντόστια. Είναι σημαντικό νορβηγικό προϊόν ο Σολομός. Τα θαλασσινά είναι το τρίτο μεγαλύτερο, 50% ε, από αυτό λαμβάνει ο Σολομός. Εμείς μόνο την Κίνα έχουμε μπροστά μας, σε ό,τι φορά την αξία των θαλασσινών που εξάγουμε. Και σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να εισαγάγει περίπου 60% των θαλασσινών που τρώτε, εμείς εξάγουμε περίπου 90%, 97% μάλιστα της 100% της παραγωγής μας. Αν δείτε την διαφάνεια αυτή θα δείτε ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει τρομακτικά τα τελευταία χρόνια και αυτό ήθελα να πω και από την αρχή σε ό,τι αφορά ειδικά την ανάπτυξη και την κοινοτομία. Υπάρχει μια εξαιρετική αλλαγή και βλέπετε πώς ε, ήταν ε, πριν από 40 χρόνια οι εγκαταστάσεις ε, και πώς είναι σήμερα. Στην Νορβηγία έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μεγάλη ακτογραμμή με μέτριο αστερμοκρασίας νερό Οπότε υπάρχουν πάρα έχει υπάρχει πάρα πολλή χώρος και πάρα πολλά σημεία για να μπουν να δημιουργηθούν τέτοιε εγκαταστάσει. Έχει όραμα η βιομηχανία μα, είναι καινοτόμα, είναι ε, σκληρά εργαζόμενοι και έχει πολλού αφουσιωμένους εργαζόμενου. Επίση, ε, θέλουμε να έχουμε την βούληση να επενδύσουμε. Είχαμε και την πολιτική υποστήριξη, βέβαια, που είναι κεφαλαίο σημασία όταν δημιουργείται μια νέα βιομηχανία σαν αυτή είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε την πολιτική υποστήριξη και όπως είδατε είμαστε μεγάλος εξαγωγέας και, σημαντικό, και ο Σολωμός είναι σημαντικός για τη χώρα. Έχουμε σαφείς, αυστηρούς κανονισμούς και πρέπει να πω ότι η δική μας βιομηχανία χρειάζεται αυστηρούς κανονισμούς και αυτό καταδείχθηκε σε άλλες χώρες. Γιατί αν ε, δεν υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί, τότε καταραίουν οι βιομηχανίε. Ε, μία από τις επιτυχίες της Νορβηγία ήταν ότι είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών θεσμών, των ρυθμιστών και της βιομηχανίας. Συνεργαστήκαμε όλοι εμείς για να δημιουργήσουμε αυτή τη βιομηχανία και βεβαίως ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά ε, Σολομού με μια ανάπτυξη της τάξης του 5-10% το χρόνο. Αν δείτε ε, μία από τις εγκαταστάσεις μας η οποία αποτελείται από αυτά τα δαχτυλίδια, θα σας, δώξω, θα σας δείξω ποιο είναι το μέγεθός τους, αλλά εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια τάση να, υπάρξει μεγαλύτερη, να υπάρξουν μεγαλύτερες ζώνες ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης με μεγάλες ε, μονάδες παραγωγής. Στην Νορβηγία προσπαθούμε να πείσουμε τους ε, συναδέλφους μας στη βιομηχανία και τις αρχές ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ακτογραμμή μας σε μεγάλες ε, ε, εκτάσεις που μπορούν να τις, που διαχειριστούμε με ολοκληρωμένο τρόπο και αυτό έχει να κάνει και με τη βιοασφάλεια και με την αποτροπή α, της εξάπλωσης ασθενειών. Γιατί σας δείχνω τώρα αυτό το ξενοδοχείο, το Ρίκα Χέν είναι το ξενοδοχείο αυτό, πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Τρόνχαϊμ. Και αν δείτε, βλέπετε, τα, αν δείτε εδώ αυτή τη διαφάνεια, ε, βλέπετε πόσο είναι το μέγεθος των δαχτυλιδιών που σας έδειχνα πριν. Μιλούμε για περίπου 160 ε, μέτρα διάμετρο και πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε αυτόν τον όγκο υπάρχει 97% ε, νερό. Δηλαδή το, τα ψάρια είναι μόλις το 3% του όγκου αυτού του τεράστιου δαχτυλιδιού ε, δίσκου. Ε, είπαμε ότι υπάρχουν αυστηροί ε, ε, κανονισμοί. Το 2006 ξεκίνησε η οθετήθηκε η πράξη για την υδατοκαλλιέργεια. Βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα για την άδεια, για τη μεταφορά, για την υποθήκευση, την καταχώρηση των αδειών υδατοκαλλιέργειας, περιφαλοντικές ανησυχίες κτλ. Η κυβέρνηση πέρσι υπέβαλε μια στρατηγική για την βιώσιμη παραγωγή. Οι βασικοί θεματικοί τομείς εδώ σχετίζονται με την ε, γενετική σύνδεση και τις, ε, την εμόλυνση, τις εκπομπές, τις ασθένειες, τη χρήση της, ε, της ζώνης και τροφές και πόροι, πηγές τροφών. Ένα από τα θέματα είναι ότι καλλιεργούμε ε, στο λαιμό του Ατλαντικού και επίσης υπάρχει και άγρος στο λαιμό του Ατλαντικού. Ε, όπως ε, είμαι σίγουρος ότι όλοι σας θα γνωρίζετε ότι ο σολομός του Ατλαντικού και τα αποθέματα του παγκοσμίω είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει και στην Νορβηγία. Παρόλο που ακόμη έχουμε αρκετό απόθεμα σε αρκετά καλή κατάσταση. Στη βιομηχανία μας λοιπόν μας κατηγόρησαν ότι είμαστε κίνδυνος για αυτά τα αποθέματα άγριου Σολομού μέσω των διαφυγών του Σολομού και της ε, ε, εξάπλωσης των ε, ασθενειών, παρα, παρασίτων κτλ. Και μπορώ να σας πω ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποτροπή της διαφυγής των ψαριών και την αντιμετώπιση των ασθενειών και των παρασίτων τα οποία μπορεί να μεταφερθούν από τα δικά μας ψάρια στα άγρια ψάρια, στον άγριο σολομό. Αυτή είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται και όπως ε, σας είπα, έχουμε επικεντρωθεί, το έχουμε θέσει ως βασική μας προτεραιότητα. Ε, προσπαθούμε να ε, ελαχιστοποιήσουμε και τις απορρίψεις από τις, από τις ώστε η, το, η ποιότητα του ύδατο και του πυθμένα να είναι καλή. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε την εξάρτηση από, την, από τις πρώτες για, τα, για τις Επίσης προσπαθούμε συνεχώς και ενεργά να εμπλέξουμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς Ξέρουμε ότι η καλλιέργεια σολαμού γίνεται στη θάλασσα που ανήκει σε όλους μας. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια είναι τα, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν ε, τη θάλασσα. Κάποια άλλα είδη καλλιέργειας θα μπορούσαν ίσως να είναι ε, παράγοντες ε, μείωσης της ποιότητας του θαλασσίου νερού. Πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν στο Παρίσι σε μια συνάντηση που ονομαζόταν η Σύνοδος Κορυφής για τις Ιχθυοτροφές. 620 ε, άνθρωποι μαζεύτηκαν για να συζητήσουν τη βιωσιμότητα των ιχθυοτροφών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο ενδιαφέρον προκαλεί. Ξέρουμε πως πολλοί από τις περιβαλλοντικές ομάδες βαθμολογούν το, τις και δίνουν στους καταναλωτές πίνακες βαθμολογίας με ποια προϊόντα ανάλογα με τη βαθμολογία να αγοράζουν και ποια όχι. Οπότε είναι κάτι που το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και εμείς υπόψη μας. Όλοι ενδιαφερόμαστε ώστε η παραγωγή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη γίνεται. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες αλυσίδες υπεραγορών ε, λένε πως ε, θα αρχίσουν να, να παρέχουν μόνο βιώσιμα ε, Το είδαμε στη ΣΥΠΑ, το, το βλέπουμε να γίνεται και στην ε, Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι προχωρούν σε ένα σύστημα εθελούσιας πιστοποίησης. Σήμερα, ας πούμε, για τα άγρια ψάρια έχουμε το Συμβούλιο, το MSE, και στις ε, υδατοκαλλιέργειες προς το παρόν έχουμε κάποια ε, περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα, αλλά προς το παρόν για, το, για την καλλιέργεια σολομού τουλάχιστον δεν έχουμε πρότυπα που να είναι αρκετά καλά σε σχέση με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Υπάρχουν κάποια πρότυπα που προσπαθούμε να εκπονήσουμε τώρα ένα από αυτά το εκπονεί η GAA, η Παγκόσμια Συμμαχία για την Αδετοκαλλιέργεια. και, και μια πάρα πολύ ε, ενδελεχής διαδικασία είναι αυτή που ε, διεξάγει το ε, Συμβούλιο της ΒΒΕΦ για τον, με το σχετικό διάλογο για την υδατοκαλλιέργεια στον οποίο και συμμετέχουμε. αυτό θα καταλήξει σε ένα νέο πρότυπο για την βιώσιμη παραγωγή σολομού Αναφέρθηκε από τον κύριο Στίβενσον ότι ο Σολομός είναι εξαιρετικός μετατροπέας ε, ηχθείοτροφών που είναι αλήθεια. Δεν έχω τώρα βέβαια το χρόνο να μπω σε όλη τη λεπτομέρεια αυτού του θέματος, αλλά στην Ορβηγία τουλάχιστον και νομίζω και σε άλλες χώρες που καλλιεργούν σολομό δεν υπάρχουν άλλα ζώα που να είναι τόσο ε, αποδοτικά σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηχθείοτροφών. Πολλέ φορές μας κατηγορούν ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά και ηχθιοτροφέ. Εμείς όμω, αντίθετα, μειώνουμε στη βιομηχανία μας τα επίπεδα ε, χρήση αυτών των ε, ουσιών. Έχουμε μειώσει την ε, χρήση των ηχθιοτροφών. Το 90 η συμπερίληψη εχθιών για, το... για τη συντροφή των Σολομών, το ήταν 65%, σήμερα είναι περίπου 25%. Και έχουμε και κάποιες, ε, κάποιες ειδικέ καλλιέργειες οι οποίες μπορεί να κατεβάσουν το ποσοστό αυτό ακόμη και στο 15%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να έχετε υπόψη σας ότι ο Σολομός ή άλλα ψάρια δεν χρειάζονται ειδικέ πρώτες χρειάζονται πρωτεΐνες, αμινοξέα, λίπαρα οξέα. Επομένως, δεν μπορούμε απλώς να μιλούμε για τις ομάδες ε, πρώτων υλών. Πρέπει να μιλούμε για συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Αν δείτε τώρα την παραγωγή ε, ηχθειοτροφών, ε, είναι λίγο πολύ ίδια τα τελευταία 30 χρόνια. Βλέπετε μια πράσινη γραμμή στο γράφημα εδώ. Βλέπετε την αύξηση της ε, παραγωγής ε, παγκοσμίως του Σολομού και βλέπετε ότι η δική μας βιομηχανία δεν είχε, κανένα, δεν, ε, δεν είχε καμία επίπτωση στην χρήση των ηχθειοτροφών. Στην Ορβηγία έχουμε προβλήματα με τη διαφυγή. Το 2004 είχαμε ένα νέο πρότυπο, υποχρεωτικό πρότυπο, και όπως βλέπετε, ε, χρειάστηκαν λίγα χρόνια πριν αρχίσει να λειτουργεί και να αποδίδει καρπούς. Και βεβαίως χρειάστηκαν και επενδύσεις της τάξης του 5, των 5 δισεκατομμυρίων. Αλλά βλέπετε ότι γύρω στο 2006 η διαφυγή μειώθηκε. Βέβαια, εντάξει, ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μα. Από, το, από το 2006, συγγνώμη. Η διαφυγή μειώθηκε. Ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μα, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι, είμαστε προς, ότι πάμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Επίση, έλεγχο ε, των ε, παρασίτων. Ίσως κάποιοι να το γνωρίζετε το παράσιτο αυτό. Και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε βιολογικά, ε, με, βιολογικά μέτρα. Υπάρχουν βέβαια τώρα κάποια είδη ψαριών τα οποία μπορούν να ουσιαστικά τρώνε αυτά τα παράσιτα από τους σολομούς. Αυτό το βλέπουμε όλο και σε περισσότερες φάρμες να συμβαίνει στην Νορβηγία. Και τώρα αρχίσαμε να καλλιεργούμε αυτά τα ε, είδη. Οπότε ε, καλλιεργούμε το ψάρι, αλλά καλλιεργούμε και το εργαλείο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παρασίτων του Σολομού. Συμμετείχαμε, δίνοντας δεδομένα, στην πρώτη παγκόσμια μελέτη που έγινε για τις εκπομπές ε, των ε, αερίων του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια ε, Σολομού. Η έρευνα αυτή έγινε το 2008-2009 και όπως βλέπετε εδώ στον πίνακα ο καλλιεργήσιμος Σολομός είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τις ε, εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, με ανέφερα και τον τομέα της έρευνας. Πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε να δημιουργούμε την πλατφόρμα για την ε, τεχνολογία και την ανάπτυξη και εκεί ε, καθορίσαμε ποιοι είναι οι κανόνες ε, που θα μας απασχολήσουν, ποιότητα και καταναλωτής, τεχνολογία και συστήματα, βιολογικός κύκλος ζωής, βιώσιμες, ε, βιώσιμες ζωοτροφές, ε, περιβαλλοντική ελοκλήρωση και υγεία των ψαριών και ευζοία. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι τομείς για τους οποίους γίνεται έρευνα ε, και το, τους παρακολουθούμε επισταμένα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν θέλετε οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες για το πώς η εταιρεία μας ε, μελετά τα θέματα βιωσιμότητας, έχετε την έκθεση από το 2008 εδώ. Ε, βλέπετε, ποια είναι, βλέπετε το σύνδεσμο και σύντομα θα υπάρξει και η έκθεση, θα δημοσιοποιηθεί και η έκθεση του 2009. Αυτή είναι η έκθεση του 2008 η οποία, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, είναι η πρώτη έκθεση τέτοιου είδους για τη δική μας βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα φοιτητών Σκοτσέζων από τη Σκοτία που κάθονται εδώ πίσω μου. Προφανώς προέρχονται από μία περιοχή που εξαρτάται πολύ από την αλία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αλίας. Συζητούμε θέματα που αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή σας, όπως είναι η δετοκαλλιέργεια και αυτή του Σολομού. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ, ανάμεσα στους βουλευτές αυτής της ε, Επιτροπής. Έχουμε σημαντικούς βουλευτές που εκπροσωπούν τη Σκοτία. Τον κύριο Χάουτον, ναι, Λοιπόν, ο κύριος Χάουτον και ο κύριος Στίβενσον εκπροσωπούν τη Σκωτία και εκπροσωπήστε άριστα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία Δον Πόρτσες, η ειδική του Marine Conservation Society του Εδιμβούργου. Καλώς ήρθατε. Εκπροσωπείτε πάλι σκοτία. Θα μιλήσει. Όλοι οι Σκοτσέζοι είναι τώρα εδώ. Σύμπτωση. Θα μιλήσει τώρα που είναι όλοι οι Σκοτσέζοι εδώ. Θα αναφερθεί και εκείνη στο ενδιαφέρον θέμα της υδατοκαλλιέργειας και έχει το λόγο για ένα τέταρτο Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσω ευχαριστώντα σα που μου δίνετε τη δυνατότητα να σα παρουσιάσω το θέμα μου μπροστά σε όλου. Είμαι η Ντόν Πέρτσις και είμαι υπεύθυνη για το καλλιέργεια στην ε, υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για, την, για τη συντήρηση τη θαλάσσια ζωή. Είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προστατεύει τα, την πανίδα τη θάλασσα. Θα ήθελα να αναφερθώ στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη. Πώς διαμορφώνεται ε, ο τομέας στο μέλλον. Ποιες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αναπτυχθεί ο τομέας βιώσιμα. Τέλος, να δούμε ποια πορεία μπορεί να πάρει ο τομέας στο μέλλον. Να κάνω κάποιες προβολές. Ο κ. Μελάνο είπε κάτι στην αρχή. Θέλω να βασιστώ σε αυτά και να αναφερθώ και στα πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή και το θέμα των ζωοτροφών που αναφέρθηκε. Θέλω να θίξω. Uh, τι μπορεί να οδηγήσει τον τομέα προς ανάπτυξη και τι προκλήσεις αντιμετωπιστούν λόγω της ανάπτυξης. Αυξάνεται η ζήτηση για τα προϊόντα της θετοκαλλιέργειας. Αυτό οφείλεται στην ε, αύξηση της κατανάλωσης κατά κεφαλή. 22 κιλά μέσος όρος είναι στην Ευρώπη και ε, από υδατοκαλλιέργειες προέρχονται τα μισά θαλασσινά. Οπότε η αύξηση της ζήτησης υποστηρίζεται κατά πολύ από την ε, παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών. Άλλος λόγος ανάπτυξης. Αυξάνεται η ζήτηση λόγω αύξησης του πληθυσμού. Άλλα δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους την επόμενη 30 ετία θα πρέπει να θρέψουμε. Όπως τα τελευταία δεκαετία πρέπει να θρέψουμε ένα δισεκατομμύριο παραπάνω ανθρώπους. Και αυτά είναι από την έκθεση του ΦΑΟ του 2006. Και βλέπετε πόσο αυξήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια η δεδοκαλλιέργεια Βλέποντας τη διαφάνεια, βλέπουμε ότι το δυναμικό δεν αυξάνεται παρκώς για να καλυφθεί η ζήτηση για τα θαλασσινά. Συνοψίζοντας λοιπόν τις συνιστώσεις ανάπτυξης Αύξηση πληθυσμού. Αύξηση κατακεφαλής κατανάλωσης. Και τα ελεύθερα αλλιεύματα έχουν φτάσει, τα αποθέματα των άγριων ψαριών έχουν φτάσει στα όρια τους όσον αφορά την εκμετάλλευση. Άρα, εξού και η αύξηση της ζήτησης από την ιδετοκαλλιέργεια για να παραχθούν τα θασανιά που θέλει να φάει ο Άρα, η παραγωγή από υδατοκαλλιέργεια πρέπει να ε, αυξηθεί με το σωστό τρόπο. Ας δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε βιωσιμότητα, τι, από τι αποτελείται η βιωσιμότητα, τι συντείνει στη βιωσιμότητα. Έχουμε πολλούς παράγοντες. Ευαισθητοποίηση, αύξηση βιωσιμότητας και εξέταση των βιολογικών συνοπιών. Οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται Θέλω να ξέρουν από πού προέρχονται όλα τα τρόφιμα, όχι μόνο τα θαλασσινά. Οι αναπολιτές πληροφορούν του καταναλωτέ για την προέλευση των θαλασσινών και γίνονται εξαρτήσει με κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει που δίνουν συμβουλέ για να ακολουθούνται καλύτερε πρακτικέ, να θαρρύνουν καλύτερε πρακτικέ. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση καταναλωτών. Σε τι οφείλεται, η ταινία The End of the Line ήταν ταινία μεγάλου μήκου που έδειχνε τις συνέπειες για την υπεραλίευση στο κοινό. Ανησυχίες για την αλία των άγριων ψαριών και την ηχθειοκαλλιέργεια των σαρκοφάγων ε, και που τη χρησιμοποιούνται ε, οι σαρδέλες για την διατροφή των ψαριών. Δημιουργήθηκε κύμα ευαισθήτων καταναλωτών που θέλουν πληροφορίε, θέλουν να διαβεβαιώσει ε, ότι θαλασσινά που τρώνε τα καλύτερα. Θέλουν να κάνουν σωστή επιλογή. Θέλουν πληροφορίε οι καταναλωτέ, να κάνουν σωστή επιλογή για βιώσιμα θαλασσινά. Και έχουμε και εμεί online πληροφορίε. Και ο προηγούμενο ομιλητή αναφέρθηκε στι πληροφορίε για του ε, οδηγού για πληροφόρηση των καταναλωτών κλπ. Και, και καρτούλες για να ξέρουν οι καταναλωτέ από πού προέρχονται τα προϊόντα και να ξέρουν τι αγοράζουν και οι λιανοπολιτές προωθούν τη βιωσιμότητα, σπρώχνουν την αγορά προς βιώσιμα θαλασσινά και το θέτουν και προς όφελός τους για την ε, αγορά και φροντίζουν τον ευαίσθητο καταναλωτή που θέλει να ξέρει που προέρχεται το θαλασσινό του. Τι θέλει ο καταναλωτής. Στην επισκόπηση του 2008 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το πώ αντιλαμβάνεται ο κόσμο την αλληλεία και τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργιών, βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Να κάποια. Υπήρχαν ανησυχίε όσον αφορά τη βιωσιμότητα των θαλασσινών. Και αυτό ήταν φραγμό για την κατανάλωση θαλασσινών. Και θέλανε και την καταθεσία για την ποιότητα των θαλασσινών που θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν κίνητρο για την αύξηση κατανάλωση. Ας δείξουμε μια ματιά στα πρότυπα πιστοποίησης. Και ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε σε τέτοια θέματα, προδιαγραφές, πιστοποίηση κλπ. και σήμανση. Να αναφερθώ κι εγώ. Πρότυπα για τη λιανική, για το λιανεμπόριο. Ανέπτυξαν δικά τους, δική του πολιτικές, δικές τους προδιαγραφές όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτού και τι προωθούν. Και ετικέτες, οργανικά πρότυπα έγινε με παρουσίαση να καλυφθεί αυτό. Θέμα σωστή διαβίωση των ζώων, οικολογική σήμανση επίση αναφέρεται. Όπω είπε και ο Πίτερ Άλισον νωρίτερα, υπάρχει και συμβούλιο για διδοκαλλιέργειε και έλεγχο. Το WWF ηγείται τη διαδικασία διαλόγου για την διδοκαλλιέργεια. Αποτέλεσμα, προδιαγραφέ, 12 προδιαγραφέ, 12 πρότυπα για διάφορα είδη υδατοκαλλιεργιών. Τα πρότυπα θα προστατεύονται από το αρμόδιο συμβούλιο. Και τα προϊόντα θα έχουν την αναγκαία σήμανση και θα ενημερώνεται ο καταναλωτή. Τα είδη θα συμπεριλαμβάνονται στα πρότυπα. Σολομό, πέστροφα, γαρίδα, ε, δίθυρα, μαλάκια κλπ. Λοιπόν, τα θέματα βιώσιμης ε, βιωσιμότητας περιβαλλοντικής να δούμε. Και ο διάλογος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή πληροφοριών. Είναι πολλά τα εμπλεκόμενα μέρη. Πολλοί που συμβάλλουν στη συζήτηση. Κάποια στοιχεία θα ήθελα να χρησιμοποιήσω από τη συζήτηση παρά να βασιστώ στις δικές μου απόψεις. Ετέσταν διάφορα θέματα. Στην ομάδα νομοθεσία, ρύθμιση, προστασία βιοτόπων, ειδών, χρήση των υδάτων, ποιότητα των υδάτων, εξωτικά είδη και χρήση τους, γενετικά τροποποιημένα οργανισμοί και χρήση τους, αντιβιωτικά και χημικά και χρησιμοποιούνται οι ασθένειε και η υγεία, έλεγχος των σαρκοβόρων και των κυνηγών που τρώνε τα άλλα είδη, ε, από πού προέρχονται τα τρόφιμα που τρέφουν τα ψάρια, τα θαλάσσια και τα χερσαία, αποδοτικότητα των ε, ζωοτροφών, χρήση της ενέργειας, κοινωνικά θέματα, ε, διαρροές, διαφυγές, επιβίωση και ανάκαμψη και ανάκτηση. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα τα καλύψει αυτά τα θέματα. Οπότε όλα τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην οικολογική σήμανση που θα χρησιμοποιείται. Να εστιαστώ σε συγκεκριμένο θέμα που απορρέει από τον κατάλογο. Ήδη αναφέρθηκε βέβαια. Ένα σημαντικό θέμα τα μεσηχή είναι η βιωσιμότητα των ζωοτροφών και η διαθεσιμότητα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση ΦΑΟ. Όσον αφορά την έκθεση για το 2006 και για το 2008 που αφορά τον τομέα. Ότι φτάσαμε στα όρια όσον αφορά την αλίευση των αγρίων ειδών από του ωκεανού και τι θάλασσε για όλα τα είδη κατανάλωση, δηλαδή και ανθρώπινη κατανάλωση και για παραγωγή ζωοτροφών για τη διδατοκαλλιέργεια. Διαθεσιμότητα πόρων αναφέρθηκε. Και πώ πρέπει να διαχέονται οι πληροφορίε. Υπό διάφορε μορφέ, την τελευταία 25 ετία η παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων έχει παραμείνει σταθερή στον αφορά τον όγκο. Και δεν μπορούμε να επεκτείνουμε για να την αλληλεία αγριών ειδών για να αυξήσουμε αυτού του πόρου. Και η βιομηχανία μεγάλωσε. Και η παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων η χρήση τους αυξήθηκε. Καινοτομία, υποκατάσταστα, καλύτερη χρήση, αύξηση ποσοστών μεταλλάξεως των τροφίμων οδήγησε σε αύξηση ε, της παραγωγής αυτών των ζωοτροφών χωρίς να πιεστούν οι πόροι. Αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή και ο τομέας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ καινοτόμοι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηχθιάλευρα και χθιέλαια με στατηγικότατο τρόπο. Ο κ. Στίβενσον αναφέρθηκε στο ποσοστό μεταπίσω των τροφίμων και τα ψάρια χρησιμοποιούνται για τρόφιμα στι ηχθειοκαλλιέργειε. Ναι, έχει βελτιωθεί ο συντελεστή, δραματικά. 1,1 στο 1 έχουμε φτάσει. Παραγωγή ηχθειοτροφών με παραγωγή ψαριών. Πόσα νοπά ψάρια χρησιμοποιούνται για να τραφούν τα άλλα τα μεγαλύτερα ψάρια, για να έχουμε το λόγο 1,1 προς 1. Αυτό που εξετάσουμε. Αναφερθήκαμε στα χθιάλευρα που παράγονται σε ένα ποσοστό 40% συμπεριλαμβάνουν ζωοτροφές. Και συμφωνώ. Αλλά και το ηχθιέλαιο χρησιμοποιείται. Και η απόδοση του ηχθιέλαιου από τον οπό ψάρι είναι περίπου 5% κατά μέσο όρο. Το φρέσκο ψάρι. Να εστιαστούμε λοιπόν και στη χρήση των ηχθιέλαιων. Είναι σημαντικό. Όπως προανέφερα, αν θέλουμε να αυξηθεί ο τομέας, χρειάζεται καινοτομία. Σημειώθηκε πρόοδος, χρειάζεται και άλλη όμως. Και ο κύριος Λαρέντο αναφέρθηκε στην χρήση των αιματαλεύρων. Ναι, είναι με πολύ καλός πόρος, αλλά υπάρχει φραγμός βιομηχανικός. Φραγμός του καταναλωτού για να χρησιμοποιηθεί το αίμα για την παραγωγή αλεύρων. Μελλοντικές εξελίξεις βασίζεται το μέλλον στην υγεία του περιβάλλοντος το οποίο κινείται και λειτουργεί. Οι καταναλωτές ξέρουν τα θέματα που αφορούν την παραγωγή των τροφίμων τους όλο και περισσότερο, όχι μόνο τα θαλασσινά. Χρειαζόμαστε οικολογική σήμανση στα προϊόντα των ηχθειοκαλλιεργιών, είναι απαραίτητο. Και χρειάζεται να έχουμε και τους αναγκαίους πόρους και θα πρέπει να έχουμε ισορροπία βιωσιμότητας και της παραγωγής των ε, θαλασσινών. Έχουν περιορισμένους πόρους, άρα για να αυξήσουμε την παραγωγή χρειάζεται καινοτομία. Και καινοτόμε λύσει όσον αφορά τι ζωοτροφέ. Καινοτόμα προϊόντα και πρακτικέ για τη διατροφή των καλλιεργουμένων ψαριών είναι απαραίτητη προπόθεση για να εξακολουθεί η ανάπτυξη του τομέα. Τονίστηκαν διάφορε δυνατότητε στην έξι Ευρωπαϊκή Ενώσεω για βιώσιμο μέλλον των υδατοκαλλιεργιών εκπονήθηκε έγγραφο το 2009. Πρέπει να γίνει έρευνα στην τεχνολογία, ούτω ώστε να γίνει η υδατοκαλλιέργεια βιώσιμη περιβαλλοντικά. Και θα πρέπει να είναι μεγάλη αξία των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, με καλή απόδοση όσον αφορά το περιβάλλον. Άρα να είμαστε σε καλύτερη θέση αυτή την παραγωγή σε σχέση με εξοκοινοτικού παραγωγού. Θέλουμε να βελτιωθεί η εικόνα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και να ανοίξουν διάφορες αγορές. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν σχετικά. Χρειάζεται να υπάρχουν πρότυπα και προδιαγραφές για περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε αυτό. Πρέπει όμως την πράξη να δούμε τι θα κάνουμε. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η οικονομία κινείται εντός του περιβάλλοντος και όχι αντίθετα προς το περιβάλλον. Κλείνοντας λοιπόν, να πω ότι πιστεύω ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν είναι φραγμός για την ανάπτυξη του τομέα. Η αύξηση του πληθυσμού και η αύξηση των καταναλωτών που έχουν μεγαλύτερη επίγνωση για το πώ παράγεται ένα βιολογικό προϊόν, μα δίνει δυνατότητα να παράγουμε υγιή προϊόντα, καλά προϊόντα, με έναν τρόπο σταθερό οικονομικά και φιλικό προ το περιβάλλον. Σα ευχαριστώ για το χρόνο σα. Να και μια φωτογραφία μου. Βλέπετε, πάω. Από πρώτο χέρι μαθαίνω τι τρέχει. Κάθε χρόνο περνάω μια εβδομάδα σε ηχθειοκαλλιέργειες για να πάρω πρώτη γεύση του πώς ε, λειτουργεί ο τομέας, να καταλάβω ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας και να δω τι μπορώ να κάνω, τι λύση να βρω για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Pues Ας περάσουμε συνεχίζοντας τον τελευταίο, θα πάρει το όλο, Δόκτωρ Πίτερ Χέφερναν του Ινστιτούτου Galloway της Ιρλανδίας, του Επιστημονικού Ινστιτούτου της Ιρλανδίας, του Galloway, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, πάντα είναι καλό στο τέλος της συνεδρίασης να είναι κανείς σύντομος, οπότε θα είμαι και εγώ σύντομος. Τα σχόλιά μου ε, αφορούν την πρόσφατη κοινοποίηση της Κομισιόν για το βιώσιμο μέλλον και τον ρόλο που έχει να παίξει η έρευνα και η καινοτομία. Ακούσαμε πολλές αναφορές να γίνονται στις προκλήσεις και στις ε, δυνατότητες που υπάρχουν το πρώτο που έχω να πω στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων που γίνονται είναι ότι αυτή η έρευνα και η κοινοτομία ε, έχει να κάνει και σε, με συνεργασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία κοινοβουλίου και κομισιών αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν ήδη. Επίσης είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο για, μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει αυτή η κοινοτομία και η ε, έρευνα. Ε, έχω μιλήσει και για την ε, νέα ε, ανάγκη που υπάρχει για, να, για την εκπόνηση μιας έρευνας, μιας πολιτικής συγγνώμη, για την θάλασσα, αλλά και για την έρευνα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ιρλανδό Ευρωβουλευτή, ο οποίο είναι εδώ μαζί μας και για τι επαφέ που είχαμε μαζί του, τον κύριο Γκάλαγκερ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων και αυτό αναφέρεται στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν, υπάρχει ανάγκη για χώρο, υπάρχει ανταγωνισμός για το χώρο, υπάρχει θέμα ε, τεχνολογιών ε, για, την για τη διαχείριση, υπάρχουν νέες, νέες τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν τα βασικά προβλήματα, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν και η, βιολο, και η βιομηχανία ε, υδατοκαλλιέργειας και άλλες θαλάσσιες βιομηχανίες ό,τι αφορά τις ε, τάσεις που υπάρχουν λόγω των κλιματικών αλλαγών. Τάσει που ε, για δεκαετίες τις είχαμε συνηθίσει μπορεί να αλλάζουν από εδώ και μπρος και είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί μπορεί να δημιουργούν και νέου κινδύνου. αλλά ταυτόχρονα μα δίνουν και νέε ευκαιρίε και πρέπει να τι κατανοήσουμε στη λεπτομέρειά τους. Γνώση ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να υποστηρίξουμε το σημείο της ε, στασιμότητας, ε, της, ε, το αδιέξοδο. Και επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις, τα εργαλεία που έχουμε για να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό που διαθέτουμε και να υποστηρίξουμε σημαντικά την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την διαχείριση και τη διοίκηση την, της βιομηχανίας. Η Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός ε, χρηματοδότης σε επίπεδο ε, καινοτομίας και έρευνας. Το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο, το έκτο, ε, επένδυσε περίπου 100 εκατομμύρια σε ευρώ σε, σε διάφορους τομείς. Μεταξύ αυτών και η υδατοκαλλιέργεια. Στο το παρόν πρόγραμμα έχει περίπου 33 εκατομμύρια. Ε, το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο. Στο παρόν πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση, υπάρχει μία αντίληψη ότι η δατοκαλλιέργεια δεν ε, αποδίδει τους απαραίτητους απαιτούμενους καρπούς έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη, να εξασφαλίσει η υποστήριξη οικονομική. Και αυτό απορρέει από τα, ε, από τα προγράμματα που υποβάλλονται ή από την έκκληση για υποβολή προγραμμάτων. Το πρόγραμμα πλαίσιο όμως επιτρέπει την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση σε κάθε τμήμα ε, της διαδικασίας. Θα σας δώσω κάποιες προτάσεις σε λίγο και συμπεράσματα, αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε στο μέλλον και θα σας το σύστηνα να με το μελετήσουμε και να κάνουμε μια κριτική αξιολόγηση. οι, κατηγορίε κατηγορίες που έχουν θεωρηθεί ως προτεραιότητες είναι αυτές που χρηματοδοτούνται, οι κρίσιμη σημασία ε, προ, ε, ε, προτεραιότητες από πολιτικής απόψεως, από οικονομικής απόψεως, από πολιτικής ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας, είναι αυτές που πρέπει για να μπορέσουμε να τις ενισχύσουμε με χρηματοδότηση. Χρησιμοποιούμε πλήρως το υπάρχον πρόγραμμα πλαίσιο για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ε, εγώ δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν χρήματα, ε, αλλά θέλω να ρωτήσω, χρησιμοποιούμε τα χρήματα που υπάρχουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Και η βιομηχανία και οι ερευνητέ λένε ότι η, ο, το ο τομέα τη ιδιωτοκαλλιέργεια προ το παρόν δεν φαίνεται να τα πηγαίνει τόσο καλά όσο θα μπορούσε στα προγράμματα που τον περιλαμβάνουν ω στοιχείο. Θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής αναφέρθηκαν από πολλού. και όντω ε, είναι υπαρκτά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έρευνα και η καινοτομία η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται για να βοηθήσουμε με αντικειμενικές απόψεις ε, όταν ε, και με στόχο την επίλυση του προβλήματος. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ευρώπη και πραγματικά είμαι πεπισμένο ότι η επιστήμη και η ε, καινοτομία θα πρέπει να υπηρετεί την ε, κοινωνία και όχι μόνο τον εαυτό τη. Η επιστήμη εδώ μπορεί πραγματικά να συμβάλλει θεαματικά με την απαιτούμενη βεβαίω υποστήριξη. Και πιστεύω επίση επειδή κάθε βιομηχανία λειτουργεί σε ένα, σε ένα περιφερειακό τοπικό επίπεδο, τοπικό επίπεδο, εθνικό και ε, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο, ότι χρειάζεται ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος μεταξύ των εργαλείων που υπάρχουν στους ε, χαράσοντες στην πολιτική, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν. Αν, υπάρχει, ε, αν υπάρξει διακοπή του συνδέσμου αυτού, τότε θα, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος ή μπορεί να επιτευχθεί εν μέρη. Οπότε δύο τα συμπεράσματα που θα σας δώσω και τέσσερις συγκεκριμένε προτάσεις για να τις μελετήσει η Επιτροπή σας. Υπάρχει ένας, ένα, μεγάλο, ένα μεγάλο αρχείο ε, ε, επιτευγμάτων στον τομέα της έρευνας και της ε, καινοτομίας. Ε, οι τεχνολογίες ανάπτυξης, η τεχνολογίες της γενετικής διαχείρισης, η τεχνολογία της υπεράκτιας ε, ανάπτυξης σε μεγαλύτερα περιβάλλοντα. Οι Ευρωπαίοι ε, ερευνητέ και οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι έχουν πραγματικά επιτύχει πάρα πολλά στη συνεργασία τους για τον τομέα αυτό και για την διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά και για την κατανόηση των ε, ωκεανών. Η Ευρώπη έχει την, ε, το επιστημονικό δυναμικό να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή. Παρ' όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι σημαντικές και για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε, η, η ένταση της έρευνας και η στοχοθέτηση της έρευνας θα πρέπει να μετακινηθούν και να περάσουν σε άλλο επίπεδο. Και αυτό νομίζω ότι το ανέφεραν πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές. Πρώτη μου σύσταση λοιπόν είναι οι ενδιαφερόμενοι ε, φορεί και αυτοί που ε, μπλέκονται στο πρόγραμμα ΦΕΜΑ και ε, όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να κάνουν μια κριτική αξιολόγηση. Οι βασικοί τομεί και τα βασικά εργαλεία είναι τα κατάλληλα και αντιμετωπίζουν επαρκώς τα θέματα που προκύπτουν με τα προγράμματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Θεωρώ ότι μια επιτροπή που ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης του προγράμματος όπως αυτή που υπάρχει για τη γεωργία η Επιτροπή ΣΚΑΡ συγκεκριμένα, αλλά μια επιτροπή που θα ασχολείται με θέματα ιδίου τύπου αλλά για την υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα αυτό και να εξασφαλίσει ότι τα βασικά θέματα αρθρώνονται σωστά και οι, προτεραιότητε κλειδιά είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Και ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, μια σωστή ολοκληρωμένη χρήση ε, των υποστηρικτικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων. Και ως προς αυτό, συχνά υπάρχουν ε, παρεκκλήσεις στους στόχους ε, της, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επιστήμη και οι κοινωνικές επιστήμες αλλά και η έρευνα μπορούν να, μπορεί να, μπορούν να βοηθήσουν στην εναρμόνιση των στόχων γιατί, έτσι ώστε να ενώσουν και τους στόχους που αφορούν τα περιβαλλοντικά και τους στόχους που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Και νομίζω ότι ο συντονισμός μπορεί να επιτύχει τον στόχο αυτό με την υποστήριξη πάντα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τρίτη μου σύσταση. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην διακυβέρνηση και στην έρευνα υποστηρίζοντας την διακυβέρνηση σε κάθε βήμα έτσι ώστε οι πολιτικές να μπορούν να ε, εκπονηθούν με βασισμένες σε, συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες αποδείξεις και δεδομένα σε κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Πρέπει να υπάρχει επίσης σαφή σύνδεσμος μεταξύ όλων αυτών. Και τέλος, να πω ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να εξετάσουμε το εξής. Επιτυγχάνουμε τον καλύτερο δυνατό σύνδεσμο μεταξύ διευθυντικών ταμείων, ερευνητικών ταμείων, περιφερειακών ταμείων και τομείων κοινοτομία για να αντιμετωπίσουμε τι κοινωνικέ πολιτικέ βιομηχανικέ ε, προκλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για όλα αυτά που μας είπαν. Έχω μία-δύο ερωτήσει. Να απευθύνω στα δύο τελευταία μέλη του πάνελ. Προς την Don Purchase. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Λέγατε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους πόρους ηχθιαλεύρων και ηχθιαλέων που χρησιμοποιούμε. Το δέχομαι, το δέχομαι αυτό. Εξετάζουμε πλήρη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και ένας από βασικούς τομείς που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο τομέας των απορρίψεων. Πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους απορρίψεων έχουμε το χρόνο. Εγώ υποψιάζομαι ότι είναι περισσότεροι. Οι μεταποιητές μου είπαν επανειλημμένα ότι θα καλωσόριζαν την εισαγωγή ενός, ε, της χρήσεως ελαίου. Να χρησιμοποιούσαν τα, τις απορρίψεις για παραγωγή χθιαλεύρων και χθιελαίων. Πώς το βλέπετε εσείς? Καλό, λογικό. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τώρα που αυξάνεται ο τομέας, αναπτύσσεται για να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση για περισσότερα εχθιάλευρα και χθιέλεα. Ο κ. Άρνεσεν ίσως. Δεν λέω τίποτα για τον τομέα της Νορβηγίας της δατολίργειας, γιατί είναι ιδιοκτήτες των δικών μας ηχθειοκαλλιεργιών στη Σκωτία, οι Νορβηγοί. Πώς τα βλέπετε εσείς, αυτό που έγινε στη Χιλή, τι δυνατότητες δημιουργούνται για μας στην Ευρώπη από αυτό που διαπιστώσατε. Ευχαριστώ. Κύριε Στίβενσον, καλώς. Να δώσω το λόγο για να απαντήσετε στον καθένα από τους ομιλητές. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Πέρτσις έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα της χρήσεως απορρίψεων για παραγωγή χθιαλεύρων και χθιαλέων Πρέπει να αποφευχθούν εν πρώτης οι απορρίψεις. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Προσπαθούμε να λαχιστοποιήσουμε ε, τις απορρίψεις μέσω ε, χρησιμοποίησης των καταλήλων εργαλείων. Χρήση τώρα των απορρίψεων στον τομέα αυτό παραγωγής ηχθιαλέων και ηχθιαλεύρων. Αν υπάρχει πολύτιμος πόρος που βγήκε από τον ωκεανό, το υπεύθυνο που είναι να το χρησιμοποιήσεις αυτό που πήρες. Αλλά τώρα τι με προβληματίζει το να χρησιμοποιούμε τις απορρίψεις. Δημιουργούμε αγορά. Εντάξει, χρησιμοποιώ μεν ότι η χρήση των απορρίψεων και η χρήση ιεσδήποτε πολύτιμης πηγής είναι κάτι πρέπει να ενθυρυνθεί και καλύτερα χρησιμοποιείται παρά να μπαίνει στις φωματερές. Απ' την άλλη όμως, μήπως δημιουργήσουμε μια ειδική αγορά για τις απορρίψεις μήπως δημιουργηθούν και ονομικά κίνητρα για τις απορρίψεις. Τι με προβληματίζει. Ένα αλλιευτικό σκάφος. Πιάνει την ποσόστοσή του ο ψαράς και έχει στον πάρει χώρο. Λέει, α, ας ρίξω ξανά τα δίχτυα μου και ας μαζέψω ό,τι να είναι. Κάποια λεφτά θα βγάλω. Η χρήση λοιπόν των απορρίψεων θα είναι κάτι καλό που μπορεί να εξεταστεί, όμως χωρίς να δίνονται οικονομικά κίνητρα για να μαζεύει κανείς επίτηδες μεγαλύτερες ποσότητες και να έχει απορρίψεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Άρνεσεν έχει το λόγο. Να απαντήσει και αυτό στην ερώτησή του. Εντάξει, καλά, με ακούτε. Θα συνεχίσω αγγλιστή. Διάλογο εκτό μικροφώνου και απάντηση στο μιλητού είναι προτιμώ τα αγγλικά. Τι έγινε στη Χιλή. Πού να σα τα λέω. Μεγάλη ιστορία, αλλά θα προσπαθώ να, τα, σας τα πω επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα, τεράστια ευκαιρία επιχειρηματική. Υπέροχε. Κατάλαβε ο κόσμος ότι υπήρχε αγορά για Σολομό. Είδαν επίσης ότι η Χιλή είχε ακτογραμμή, ένα κομμάτι της χειλή είχε ακτογραμμή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτροφή σολόμου η νότια χιλή. Υπέροχη για αυτή τη δουλειά, για παραγωγή σολομού. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε βιολογικές πτυχές και βιολογική ασφάλεια και τα συναφή μέτρα. Οι εκμεταλλεύσεις ήταν πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά και έλειπε, τι να πω, οι νόμοι δεν ήταν αρκετά αυστηροί. Και δεν επιβαλόταν ο νόμος. Δεν επιβαλόταν με αυστηρότητα ο νόμος. Δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή στη δυνατότητα να αντέξει το περιβάλλον. Πάρα πολλά ψάρια σε πολύ μικρό χώρο μαζεύτηκαν. Όταν ξέσπασε αυτή η ασθένεια, η μεταδοτική ανεμία του Σολομού, όταν συνέβη αυτό το 2007, μία από τις δικές μας εκμεταλλεύσεις ήταν η πρώτη που ανακάλυψε αυτή την ασθένεια, ο τομέας δεν ήταν έτοιμος για μία ασθένεια τόσο κολλητική, όπως η ISA, όπως είναι τα αρχικά της ασθένειας που σας ανέφερα, της ανεμίας του Σολομού, της μεταδοτικής. Η ISA λοιπόν είναι ασθένεια που διαπιστώθηκε σε Νορβηγία, Σκοτία, νήσους Φερόες και ανατολικές ακτές του Καναδά. Δεν είναι άγνωστη η ασθένεια. Είναι μια ασθένεια που μάθαμε να τη δεχόμαστε και να συμβιώνουμε. Εξακολουθεί να υπάρχει στην Νορβηγία αυτή η ασθένεια. Έχουμε κάποια κρούσματα κάθε χρόνο αλλά πρέπει ο τομέας να είναι οργανωμένος και σχεδιασμένος το τρόπος ούτως ώστε να αποφεύγει τη διάδοση της ασθενείας με τον τρόπο που διαδόθηκε στη Χιλή. Αυτή είναι η σύντομη εκδοχή της ιστορίας. Μπορώ να σας δώσω και την πλήρη περιγραφή αν έχετε χρόνο. Σας ευχαριστώ για την ώρα. Μας αρκούν αυτά. Ο κύριος Γκάρεκ έχει το λόγο. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Άρνεσεν. Οι συνθήκες πρόσβασης στην κοινοτική αγορά για το Σολομό της Νορβηγίας και τα τέλη, τα πιο ε, υψηλά τέλη που εισπράττονται όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα. Ποια είναι η άποψή του για όλα αυτά. Δεύτερον, διαδικαστικά πού βρισκόμαστε αντι και κατά των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τον νορβηγικό Σολομό. Έληξε αυτή η ιστορία ή έχει ανησυχίες ακόμα η ειχε ανησυχιες ακομα Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Τέλος, μιλήσατε για το μικρό ίχνος άνθρακα όσον αφορά την παραγωγή, την νορβηγική. Ναι. Όσον αφορά το ίχνος του άνθρακα, τι γίνεται με το σολομό που παράγεται στην Ορβηγία, που στέλνεται στην Κίνα και εκεί μεταποιείται σε φιλέτα και επανεισάγεται στην Ευρώπη. Είναι λογικό αυτό. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματά μου, κύριε Άρνεσεν. Ευχαριστώ. Κύριε Άρνεσεν. Um, let me take the last... Να απαντήσω πρώτα στο τελευταίο για το ανθρωπικό αποτύπωμα και την εξαγωγή ε, ψαριών στην Κίνα. Για τον τομέα αυτό, την αλήθεια να σας πω, δεν ξέρω πολλά, αλλά πόσο ξέρω, εάν οι ποσότητες είναι αρκετά υψηλές και μεταφέρονται ως εκατεψυγμένα ψάρια, τότε οι εκπομπές άνθρακα δεν είναι όσο άσχημες τα νόμιζε κανεί. Χωρίς όμως να έχω και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία να σας δώσω. Τώρα, για την ε, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και το θέμα του dumping. Ε, δεν θα έπρεπε να ρωτάτε εμένα για το θέμα αυτό. Και πάλι από όσο ξέρω, προς το παρόν, εξάγουμε χωρίς κανένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λεβίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Έχουμε εδώ έναν ε, ε, κύριο από γειτονική χώρα και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, το σχόλιο της κυρίας Πέρτσιος. Μιλάμε όντως για διαφορετικά πράγματα όταν μιλούμε για τα διάφορα είδη ψαριών. Είναι κρίμα που ο κύριος Άρνεσεν ε, απέφυγε το ερώτημα για, το, για τα αριθμητικά στοιχεία που του ζητήσαμε ε, για, την, ε, ε, για, το, για ποσά του, τις ποσότητες λόγω που παράγονται και είπαμε ότι το, τα περιθώρια είναι δύο προς ένα αντί για ένα προς ένα αλλά όντως μιλούμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Και ποια είναι η, αναλογία των ε, τροφών που προέρχονται από, θαλάσσιους, ε, από θαλάσσιες πηγές. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πόσα άγρια ψάρια χρησιμοποιούνται ως ε, τμήμα της, ως ποσοστό ας πούμε του παραγόμενου σολομού. Αν ας πούμε δούμε τις ζωτροφές για τις καλλιέργειες. Πώς ξέρετε ότι, αυτό το, ότι η ζωτροφή δεν προέρχεται από απειλούμενα είδη από θέματα. Η Σουηδική τηλεόραση έκανε πραγματικά ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που το ονόμαζαν Pink Gold. Πρέπει να το είδατε κι εσείς στην Νορβηγία και έλεγε ότι ε, το σαφρίδι που είναι ένα ε, ε, ψάρι με υψηλό σε που μπορούμε να το φάμε και εμείς λαμβάνεται από την Ισλανδία και πηγαίνει ως, ως ηχθειοτροφή για την παραγωγή στην, σολομού στην Νορβηγία. Το ίδιο συμβαίνει και με το προσφυγάκι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Απλώς θέλω να τονίσω στην Επιτροπή πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε περί τίνος μιλούμε κάθε φορά. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια θέματα ηχθειοτροφών, οικοεπισήμανσης, ε, πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι διατροφές. Πρέπει να ξέρουμε ότι προέρχονται από βιώσιμο υγιές απόθεμα. Μετά έχουμε και τις διαρροές, τις ε, διαφυγές από τις ε, φάρμες τις νορβηγικές. Είναι καλό που έχουν πέσει τόσο πολύ τα ποσοστά. Μιλούμε για ένα εκατομμύριο ψάρια τα οποία διέφυγαν το 2006 και πέρσι είχαν φτάσει στις 170.000. Αλλά παρόλα αυτά είναι υψηλό το ποσό και αποτελεί πρόβλημα τουλάχιστον για τα αγρία αποθέματα, για τα αποθέματα άγριων ψαριών. Είναι σημαντικό λοιπόν το πρόβλημα με το, σολο, με το σολομό. Και μετά επιπλέον έχουμε και τις ασθένειες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν ασθένειες που ε, ε, ε, μολύνουν τα αποθέματα στην Ορβηγία και στη θάλασσα και στις φάρμες. Ίσως οι καταναλωτές να θεωρούν ότι τα καλλιεργούμενα ψάρια είναι καλά γιατί βοηθούν τα άγρια ψάρια, αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά στην πραγματικότητα. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε την, ε, σε μεγάλο εύρο στην καλλιέργεια Σολομού στην Ορβηγία και παρόλα αυτά τα προστατευόμενα φιόρτ που προστατεύονται από τις, ε, από τις, ε, από τις έχουν τεράστιες διαφυγές ψαριών που ξεφεύγουν από τις ε, φάρμες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα νέα είδη που καλλιεργούνται ή που τέλος πάντων γίνονται κάποιοι πειραματισμοί. Ας πούμε καλλιέργεια γάδου. Μειώσαμε τη χρήση αντιβιωτικών στις ε, ε φάρμες ήδη πριν από 20 χρόνια. Αλλά αυτό ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει για τις φάρμες ε, γάδου. Ε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι φάρμες γάδου. Και ένα ερώτημα για την κυρία Πέρτσες. Εσείς τι πιστεύετε για το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το δυναμικό για την καλλιέργεια φυτοφάγων ψαριών Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα ε, να αναπτυχθούμε και στον τομέα αυτό. Κάποια ε, είδη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως, ή να καλλιεργηθούν ως φυτοφάγα. Ε, θεωρείτε ότι για την Ευρώπη, ας πούμε, τουλάχιστον από πλευρά περιβαλλοντικής θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θέλετε να απαντήσω στα αγγλικά ή στα νορβηγικά. Όχι, όχι. Μπορείτε ισπανικά και αγγλικά. Όχι νορβηγικά, δεν υπάρχει διερμηνία από τα νορβηγικά. Ε, λοιπόν, υπάρχει... Ε, δεν υπάρχουν τα νορβηγικά. Θα μιλήσω αγγλικά, λέει ισπανικά ο μιλητής. Λοιπόν, καταρχάς, πόσα ε, νοπά ψάρια χρησιμοποιούμε, φέσκα ψάρια χρησιμοποιούμε Το υπολόγισα τις περασμένες. 2,4 για την ορβηγική παραγωγή. Τόσο φρέσκο ψάρι χρησιμοποιείται. Βάση του χθιελαίου το απαιτουμένο. Αν υπολόγιζα μόνο τις πρωτεΐνες, άντε κοντά στο ένα θα ήμουν. Αλλά εφόσον χρειαζόμαστε ένα ποσοστό ηχθιελαίου, φτάνω στο 2,4. Αν μειώσω το ηχθιέλαιο, Μπορώ να πω και πιο χαμηλά. Τώρα όσον αφορά αυτό το στοιχείο, εγώ που εστιάζομαι, που εστιαζόμαστε εμείς στη Marine Harvest, βιωσιμότητα των αλλιευμάτων, τη βιωσιμότητα του τόπου προέλευσης των ψαριών αυτών. Εμείς θέλουμε να έχουμε βιώσιμες πηγές ηχθιελαίων και ηχθιαλεύρων. Εκεί κάνουμε προσπάθειες. Ένα κομμάτι της δουλειάς, μία αρχή, έγινε από τη Διεθνή Οργάνωση Ηχθιαλέων και Ηχθιαλεύρων, Ήχθο. Έχει ετοιμάσει νέα πρότυπα για υπεύθυνη παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιαλέων. Η μέθοδος αυτή πήρε την πρώτη πιστοποίηση. Ο μεγαλύτερο παραγωγός του Περού πήρε αυτή την πιστοποίηση. Αυτό μας ενθαρρύνει. Προσπαθούμε να σπρώξουμε πιο πέρα την αλυσίδα προς καλύτερη ε, αξία. Θα έχουμε στο μέλλον διαθέσιμο ε, ηχθιάλευρο με πιστοποίηση MSE. Όσον αφορά τον ε, Ισλανδικό βακαλάο, εγώ δεν θα σχολιάσω τις αλληλευτικές πολιτικές. Πολύ, πολύ μικρό ποσοστό αυτό του μπακαλιάρου μπήκε στην ε, εκθειοτροφή μας διότι δεν ήταν καλή η ποιότητα. Είχε το ψάρι μέσα ήδη πολύ ε, ζωοτροφή στα, στα εντόστια του, στα έντερά του και δεν ήταν καλή η ποιότητα. Πού κατέληξε? Σε τροφή για τις κότες. Και τότε εκεί μπορεί να τεθούν θέματα βιωσιμότητα. σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι. Όσον αφορά τα άλλα είδη, για το προσφυγάκι, εντάξει μειώθηκαν οι ποσοστώσεις τώρα, αλλά εστιαζόμαστε πολύ σε αυτά τα θέματα. Δεν θέλουμε να συνδεόμαστε με σκούπισμα, σάρωση των θαλασσών. Θέλουμε βιώσιμη πρώτη ύλη, είτε προέρχεται από τις θάλασσες, είτε από την ξηρά. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε. Αναφέρθηκατε στις διαφυγές. Εμένας δεν μας ικανοποιεί αυτό που μας το σκάνει τα ψάρια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρουμε ότι σχετίζεται με την ποιότητα του εξοπλισμού και με την οτροπία των ανθρώπων. Και βεβαίως γι' αυτό στην εταιρεία μας εισάγουμε γενικά, γενικές διαδικασίες πρότυπα για να αποφύγουμε τις ασθένειες, συγγνώμη διότι ο να εμποδίσουμε τις διαφυγές. Όσον αφορά αυτό το θέμα των αποδράσεων, δεν θέλω να μπω σε γενετικά θέματα, όσον αφορά τα, τα ψάρια που αποδρούν, διότι δεν είναι προφανές ότι αυτό έχει γενετική συνέπεια. Δεν αλλάζουν τα γονίδια των ψαριών, τα ίδια γονίδια είναι. Ο Σολομός της Νορβηγίας βασίζεται σε 40 άγρια είδη. Τα γονίδια είναι τα ίδια. Η συχνότητα όμως μπορεί να αλλάξει. Αυτό όπως επικίνδυνο είναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Οι ερευνητές ακόμα το ψάχνουν. Οι ασθένειες. Στην Νορβηγία έχουμε πολύ λίγες ασθένειες στα ψάρια μας. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα αντιβιωτικό σχεδόν. Είμαστε κοντά στο μηδέν. Όσο πιο κοντά στο μηδέν γίνεται. Έχουμε προβλήματα με τις θαλάσσιες, τις θαλασσόψυρες. Και ίσως να μεταπη... μεταπηδούν στα άλλα ψάρια αυτές οι ψήρες. δεν έχουμε σωστή τεκμηρίωση. Αλλά πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και να κάνουμε ό,τι μπορεί για να αποφύγουμε μετάδοση θαλασσόψυρας από τα δικά μας ψάρια στα άγρια ψάρια. Ο Ρήνος ποταμός ήταν ο καλύτερος ποταμός για Σολομό στην Ευρώπη εδώ και 100 χρόνια. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν πολλοί Σολομοί τώρα στον ποταμό Ρήνο σήμερα και δεν υπάρχουν και πολλές ηχθειοκαλλιέργειες στο Ρήνο σήμερα για πολλούς λόγους ε, είναι σε κακή κατάσταση τα αποθέματα του Σολομού. Ναι, ήδη. Τι να πω. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Στο Βακαλάο και εμείς όταν ανατήσαμε το Σολομό είχαμε προβλήματα. Θα υπάρξουν προκλήσεις προς αντιμετώπιση και επίλυση. Δεν είμαι ειδικό όμως όσον αφορά την καλλιέργεια του μπακαλιάρου, άρα δεν θέλω να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Πέρτσες θέλει να απαντήσει, θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα ίσως και μετά να απαντήσει. Ε, ε, Ευχαριστώ. Μου απευθύνεται ένα ερώτημα για συγκεκριμένα είδη ψαριών Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Στίβενσον για τον ε, ρυθμό ε, μετατροπής για, τα, για τις για το ένα προς ένα. αλλά είναι το βάρος των νοπών ψαριών που χρησιμοποιείται για να παράξει αυτό το 1,1 κιλό. Οπότε μάλλον η δική μου δουλειά βασίζεται στο να εξασφαλίσω ότι αυτά τα νοπά ψάρια είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμα και να εξασφαλίσω ότι οτιδήποτε, οποιοδήποτε ψάρι χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε ε, ε, είδος, σε οποιοδήποτε ρυθμό μετατροπής να, είναι, να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο, με τον πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτός είναι, αυτή είναι η βασική μου δουλειά. Και επίσης επικεντρώνομαι στο πώς μπορούμε να βρούμε εναλλακτικά συστατικά ε, τροφής για να ενισχύσουμε ή να ε, εμπλουτίσουμε τα θαλασσιά συστατικά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι κύκλοι ζωής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την, ε, τα ψάρια αυτά με βιώσιμο τρόπο και να απαντήσω στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι η ε, καλλιέργεια ε, των φυτοφάγων ψαριών είναι χρήσιμη φυσικά. Η τηλάπια ας πούμε. Υπάρχει κάτι καλλιέργεια τηλάπια στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με σε πολύ συντονισμένο σύστημα και υπάρχει και αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο για το συγκεκριμένο είδος. Παρόλο που μιλώντα με του λιανοπολιτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθούν να ενισχύσουν και να πουλήσουν αυτό το ψάρι, αυτό το είδο, υπάρχει μεγάλο φράγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ευρώπη, να πιστεί ο κόσμο να το καταναλώσει αυτό το ψάρι. Και εκεί ίσω αυτό είναι ένα τομέα έρευνα που θα μπορούσαμε να δράσουμε. Και εκεί θα μπορούσαμε και εμεί ω οργανισμό να δράσουμε, να προσπαθήσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε γνωστούς σεφ να, για να μαγειρέψουν, να, να φτιάξουν κάποια μενού με το συγκεκριμένο ψάρι, ώστε να, έτσι να κινηθεί λιγάκι το ενδιαφέρον των πολιτών. Επίσης, ο Κυπρίνος είναι ένα πολύ ε, καλό ψάρι και θα μπορούσε να, να καλλιεργηθεί και ως φυτοφάγο, αλλά κανένας δεν θέλει να φάει Κυπρίνο τελικά, όπως είδαμε. Ο κύριος Γκάλαγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώ ε, δεν μπόρεσα να είμαι εδώ από την αρχή με διάφορε παράλληλε συνεδριάσει που τρέχουν, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσω να τι διαβάσω αργότερα. Σε σχέση με τι απορρίψει, θα πω απλώ ότι Φυσικά αντιτιθέμεθα πλήρω στι απορρίψει. Δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τι απορρίψει. Μπορούμε να ε, ποσοτικοποιήσουμε τι φορτώσει, τι εκφορτώσει, αλλά όχι τι ρίχνεται πίσω στη θάλασσα. Και σε αυτά που εκφορτώνονται θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν για κάποιου στόχου που θα είναι ε, άλλοι στόχοι εκτό του να πάνε να γίνουν ζωοτροφή. Και νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μα θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, με τι απορρίψει, σε συνεργασία με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ όσου εμπλέκονται στο τομέα της γεωργίας. Η, είναι πάρα πολύ γνωστή στην α, Ιρλανδία και εντάξει υπήρξαν διαφορέ που είχαμε αντίθετε απόψεις για τι τιμέ, για τι ελάχιστε τιμέ των εισαγωγών κτλ. Αλλά πραγματικά όλοι εκτιμούμε πάρα πολύ τη δουλειά σας. Και είναι μια, ένας τομέας με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Υπάρχουν, υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ε, όντως επειδή ακριβώς είναι υψηλού κινδύνου. Γιατί υπάρχουν και πολλές φορές προβλήματα, δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Αλλά υπάρχει και θέμα με όσους ανθρώπους χάνουν ε, την θέση εργασία τους, χάνουν τη δουλειά τους. Και όσο, μπορούμε, όσο περισσότερο μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή, αυτή την, αυτό τον τομέα και την, ε, το, και την τοποθεσία στην οποία καλλιεργούνται τα ψάρια, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Όταν κανείς σκέφτεται την ιδιωτοκαλλιέργεια, σκέφτεται σολομό. Αλλά τα πράγματα ξεπερνούν το σολομό. Το θέμα είναι να έχουμε τις ευκαιρίες για ανάπτυξη είτε θα είναι ε, των καλλιεργειών ε, είτε είναι ε, καλλιέργεια θηνοειδών είτε είναι άλλα είδη ψαριών. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της έρευνας. Μερικές φορές δεν συνδέουμε την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία με τα ψάρια, αλλά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εκεί και ο Πίτερ Χέφνερ ε, πραγματικά έχουν ασχοληθεί εντατικά με αυτό και φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε ασχοληθεί για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν επαρκή κονδύλια για τον τομέα αυτό. Οπότε η έρευνα είναι σημαντική για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερα είδη καλλιεργούμενων ψαριών εκεί που είναι σημαντικό για αυτούς που επενδύουν γιατί είναι εξίσου σημαντικό και για αυτούς που ε, χρειάζονται την ε, θέση εργασίας που τους προσφέρει αυτός ο τομέας. Η κυρία Πέρτσες. Uh, uh, Γενικό σχόλιο είναι αυτό και όχι ερώτηση. Πολλά υπόθηκαν το απόγευμα. Πόροι για την έρευνα εθίγησαν. Το υποστηρίζω αυτό, χρειάζονται χρήματα. Όμως, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στο επόμενο βήμα. Τι γίνεται μετά την έρευνα. Έγινε πάρα πολύ έρευνα και πολυτιμότατη εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στην Ορβηγία. Πρέπει να θυμόμαστε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η έρευνα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το να πάρουμε πόρους από την έρευνα και από τις δοκιμές και να χρηματοδοτούμε τις ιδέες που θα μπουν σε εμπορικές δοκιμές. Αυτό θέλουμε. Εμπορική δοκιμή, πειράματα που θα δείχνουν ότι οι καινοτόμες πρακτικές, οι καινοτόμες ζωοτροφές, οι καινοτόμες παραγωγικές μέθοδοι πράγματι μπορούν να παραγάγουν υγιή θαλασσινά φιλικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με βιώσιμο τρόπο. Που πουλιέται, έχει αξία, που αρέσει τον καταναλωτή, το τρώει καταναλωτής. Τι θέλω να πω. Καλή και άγια η έρευνα θέλει χρήματα, αλλά πρέπει να δώσουμε χρήματα τόσο ώστε η έρευνα να εφαρμόζεται, να βρει πρακτικές λύσεις και να παράγουμε είδη τα οποία να μπορούν να απολούνται και να ενθαρρύνουμε του καταναλωτές να τα τρώνε. Eh, Ο κ. Κουεφ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ που διοργανώσατε κυρία Πρόεδρε αυτή την ανταλλαγή απόψεων άκρως ενδιαφέρουσα που, που παρατείνει θα έλεγα τη συζήτηση που διεξήχθη ε, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί βιωσίμου που πετέλεσε αντικείμενο εκθέσεως του κυρίου Μιλάνα που είναι παρόν. Θεωρώ, για να είμαι λακωνικός, ότι τα μαθήματα που αντιλούμε από την ανταλλαγή είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, η πρόκληση όσον αφορά το βιώσιμο χαρακτήρα της υδατοκαλλιέργειας τίθεται όσον αφορά την εντατική υδατοκαλλιέργεια. Η εκτατική υδατοκαλλιέργεια που ανέφερε ο κ. Γκάλαγκερ προηγουμένως δεν αντιπροσωπεύεται αυτή κάθε αυτή και λυπούμεθα για την απουσία ε, των εκπροσώπων της. Και δεν εκπροσωπείται και ο τομέας της εκτατικής καλλιέργειας όπως παραγωγή κυπρίνου και άλλων συναφών ειδών. Διότι η βιωσιμότητα αυτών των δραστηριοτήτων δεν τίθεται με παρόμοιο τρόπο όπως αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Τώρα, όσο, όσον αφορά τις παρεμβάσεις της βιομηχανίας, ε, του τομέα μάλλον και τις συστάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα. Αναγνωρίζει, όπως και ο τομέας άλλωστε, ότι πράγματι καταρχάς υπάρχει πρόβλημα χωρικών εντοπίσιμων ίσως όχι, όχι μόνο εις Νορβηγία αλλά και εις Νότων για την ανάπτυξη της ειδοκαλλιεργίας και είναι παράγον αποφασιστικό για την ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή θετοκαλλιέργεια. Δεν υπάρχει επαρκή χώρο. Οι τοπικέ κοινότητε, περιφερειακέ δεν δίνουν και άλλε άδειε που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη τη ειδοκαλλιεργία, ούτε θαλασσία τιάφτη, ούτε ποτάμια. Είναι γεγονό προφανές που εμποδίζει την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Δεύτερη παρατήρηση που εξέφρασε ο τομέα αφορά την νομιμότητα, η ισότητα μάλλον της ντόπια παραγωγής έναντι των εισαγωγών. Και εμείς το εξετάσαμε αυτό και συμπεριλάβαμε ότι δεν υπάρχει στρέβλος στον ανταγωνισμό πλευράς υγειονομικής από τη στιγμή που διεξάγονται με σωστό τρόπο οι έλεγχοι. Και όσον αφορά το περιβάλλον, ε, υπήρχαν διαφορές νομοθετικές θεσίας μεταξύ κοινοτική νομοθεσίας και νομοθεσίας τρίτων χώρων. Αλλά υπήρχε ένα gap, ένα κενό μεγάλο, σημαντικό. Και υπήρξε και τρίτη παρατήρηση. Περί του διοικητικού άχθους και του χρόνου που χρειάζεται την αδειοδότηση. Δεν υπάρχει αδειοδότηση, δεν υπάρχει άδεια, αλλά αν υπήρχε θα χρειαζόταν τόσος χρόνος να χορηγηθεί που αυτό θα ακινητοποιούσε την ε, υδατοκαλλιέργεια. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την όλη ανάλυση. Συμφωνεί επίσης με την ανάγκη εξέτασης μέτρων για να μειωθούν οι συνέπειες όλων αυτών που προαναφέρθηκαν. Όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η αρμοδιότης όσον αφορά τον τομέα της ιατροκαλλιέργειας δεν είναι ε, ισχυρή κοινοτική αρμοδιότης αλλά δύναμη μαζί με τα κάτι μέλη και τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες, την τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τα θέματα τα χωροταξικά εκεί θα πρέπει να εξαχθούν συζητήσεις. Τέλος, όσον αφορά τις ανταλλαγές για, τα, για τις απορρίψεις. Την πολιτική περί απορρίψεων είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε εδώ, όμως είναι αμφισβητήσιμο ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε την περίσταση οι αλληλείς οι ίδιοι να αναπτύξουν μια αγορά απορρίψεων μία απορριμμένων ψαριών που θα τα διαφορετικά. Δεν υπάρχουν τα κίνητρα για τα ψάρια που πηγαίνουν για παραγωγή χθιαλεύρων. Σήμερα τουλάχιστον. Αυτό είναι κάτι που συνδέεται με την ε, πολιτική που ακολουθείτε για την διατροφή και νομίζω ότι στις 3 Μαρτίου θα διεξαχθεί εκ νέου μια ανταλλαγή από αυτών των θεμάτων εφόσον ε, το Κοινοβούλιο διοργανώνει μία συνεδρίαση που αφιερώνεται αποκλειστικά στην διατροφή εκείνες τις μέρες. Ευχαριστώ και για να κλείσουμε ο κύριος ο εισηγητής μας, ο κύριος Μιλάνο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός, επιγραμματικός, σύντομος. Ευχαριστώ όλους η συζήτηση υπήρξε άκρως ενδιαφέρουσα. Και από πλευράς εμπειρογνωμόνων που ακούστηκαν και από πλευράς παρεμβάσεων των συναδέλφων μας, βουλευτών, που με βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τις τοποθετήσεις του καθενός από εμάς όσον αφορά το ζήτημα. Πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα της διατάξεως του κανονισμού, της συντάξεως του κανονισμού. Οι παρεμβάσεις έδειξαν ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο προβληματισμού συγκεκριμένο σε αυτή την Επιτροπή. Όσον αφορά την γνωμοδότηση επί τη ανακοινώσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπερβλήθη στο Κοινοβούλιο. Και μπορούμε να σταματήσουμε ένα στάδιο πριν, ένα λεπτάκι πριν από αυτό το στάδιο. Δεν το λέω αυτό διότι. Μάλλον το λέω για να αποφύγουμε να μπούμε στι τεχνικέ λεπτομέρειε που αφήνει πολύ λίγο χώρο στη διαμόρφωση πολιτική. Ας πάμε στις πολιτικές επιλογές που θα πρέπει να γίνονται τώρα. Έχουμε ένα δεδομένο. Μια αγορά που αναπτύσσεται. Καταναλωτές που ζητούν, έχουν απαιτήσει και μια απέτηση όλου του πλανήτη που ζητά ε, διατροφή, τρόφιμα, παραγωγή τροφίμων και όλα αυτά οδηγούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Από κάποιου κάποιος θα παράγει προϊόντα υδατοκαλλιέργεια. ψάρια από υδατοκαλλιέργεια. Εγώ πιστεύω ότι προϊόντα εντός συγκεκριμένων κανόνων και συστημάτων ελέγχου για σκοπό αυτό για να παράγει τα προϊόντα που χρειάζεται ο, ο πλανήτης αλλά χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Καλύτερα να παράγουμε εδώ με κανόνες παρά Από εκεί ξεκινώ, αυτή την προϋπόθεση. Τώρα, πότε, πώς. Εμείς έχουμε ακτές πάρα πολλές Έχουμε πάρα πολλούς κατοίκους επίσης και μια κατανάλωση προσμετρήσιμη στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να βρούμε το σωστό τύπο που θα είναι η ισορροπία. Άρα μεταξύ ακτής, χιλιόγραμμα παραγωγής και κατοίκους. Αυτό θα μπει στην εξίσωση. Όταν μας λένε μέχρι πού, μέχρι πότε, Ποιο θα είναι ο στόχος. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι συμβατό. Γι' αυτό εγώ δεν θα περίπτα την πρόταση που έκανα στην αρχή. Το σχεδιασμό το χωροταξικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν μιλάμε για χωροταξία της θάλασσας, τι εννοούμε. Πολεοδομία της θάλασσας, χωροταξία της θάλασσας. Θέλουμε εντός ενός πλαισίου συγκεκριμένου να κάνουμε κάτι. Ίσως στη Γαλλικία να βρέθηκε, να βρέθηκε το σωστό πεδίο ισορροπίας έκταση ακτών, χιλιόγραμμα, κάτοικοι. Υπάρχουν άλλοι, ε, άλλες περιοχές που δεν υπάρχει αυτή η συμβατότητα και αυτή η ισορροπία. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πηγές. Δεν μπορούν τυχαία να μοιραστούν. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τη χρήση των πόρων συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης αντί άλλου. Η χρήση του το τρόπο των πόρων μπορεί να οδηγήσει συμβατότητα με τους περιβαλλοντικούς όρους και συνθήκες. Βέβαια, υπό την προπόθεση υπάρχει χώρος. Ήδη σχεδιασμός ο τωρινός μπορεί να παράγει καλύτερα. Μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Σχεδιασμός, λοιπόν. Σχέση κατοίκων, εδαφών, ακτών παραγωγής μεγαλύτερη αξιολόγηση των υπαρχόντων στοιχείων, πιο βιώσιμη προσέγγιση, να είμαστε πιο παραγωγικοί με αυτά που έχουμε. Για τις αγωγές, αυτές έχουν άμεσες συνέπειες. Αν ένας κανονισμός προωθεί αυστηρές συμπεριφορές και απαιτεί εχέγγυα διάφορα, πολιτική, σημάτων, φερρυπίν, τι είναι βιώσιμο, τι είναι βιολογικό να αναφέρεται στην ετικέτα. Αν υπάρχει συνέπεια, χωρίς να δημιουργήσουμε τελωνιακούς φραγμούς, αυτός μπορεί να γίνει ένας μηχανισμός που θέτει τροχοπέδι στις αγωγές. Και θα πρέπει τα εισαγόμενα προϊόντα να ταιριάζουν καλύτερα στις προδιαγραφές των αγορών μας. Στο τελευταίο που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ότι δεν είναι κοινοτικό ζήτημα. Ίσως τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ίσως αυτό είναι κάτι, ξέρω εγώ, δεν θα πρέπει να κάνουμε αθλητικού τύπου εκδηλώσεις. Πρέπει να κάνουμε προβληματισμό εδώ πολιτικό. Δεν βγάλουμε αθλητικές εκδηλώσεις. Όταν καταφτάνει μια έκθεση στο κοινοβούλιο, δίδεται μια εντολή. Είναι αντικείμενο σε αυτή η έκθεση. Και από πλευρά Συμβουλίου πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει η Ευρώπη να αξιολογήσει κάποια πράγματα. Και θέματα ίσως που αφορούν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Αν πούμε ότι η ανακοίνωση του 2002 ήταν αναποτελεσματική όσον αφορά όλα αυτά που ετίθενται, απλούστευση, εναρμόνιση, ταχύτητα, διαδικασιών, του συστήματος. Αν το λέγαμε αυτό εδώ και κάποια χρόνια, βλέπαμε έναν κόσμο πήγαινε σε μια κατε... Ε, κατεύθυνση και εμείς σταματήσαμε. Τι γίνεται. Ανησυχώ. Ετοιμάζουμε στατιστικές, κάνουμε ανάλυση. Και είπαμε ότι ο κόσμος αναπτύχθηκε πολύ, εμείς λίγο, ένα προς έξι κλπ. Αν δούμε τα στοιχεία του Σολομού μόνο, όπως αναφέρθηκε, η μόνη αύξηση βλέπουμε αύξηση του Σολομού και μία μείωση των υπολείπων, αν είναι σωστά τα στοιχεία. Διότι ποτέ δεν αναλύσαμε τα στοιχεία κατά οικογένειες ειδών. Άρα τίθεται και το θέμα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων των άλλων. Αυξήθηκε έναντι των άλλων ειδών ο Σολομός, τα άλλα λευκά ψάρια της Μεσογείου και των διαφόρων οστράκων, μαλακίων κλπ. Εκεί είχαν μείωση τα άλλα είδη, τα άλλα θαλασσινά. Είναι πολύ επικαιρό το θέμα. Άρα πρέπει να ασχοληθούμε τι γίνεται από τα διάφορα είδη. Τέλος, το θέμα των τροφίμων θέλαμε ότι ήταν των τροφών ήταν περίπλοκο. Περίπλοκο ποσοτικά και ποιοτικά. Και όσον αφορά το συσχετισμό το ψάρι τρώει το άλλο, το ένα ψάρι τρώει το άλλο και ποια είναι η αναλογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους σας. Δέα λοιπόν αυτό για τους Κυπρίνους που διατρέφονται για να τρέφονται τα σαρκοβόρα ψάρια. Τρέλη ιδέα είναι αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μιλάνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο για τη συμμετοχή του σε αυτή την ακρόαση και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για όλους μας και θα σκεφτούμε, θα τα λάβει υπόψη ο κύριος Μιλάνα και θα τα λάβει υπόψη την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε αυτό το σημείο και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα, οπότε πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά τις αποφάσεις που υιοθέτησαν οι συντονιστές. Ε, πιστεύω ότι όλες οι αποφάσεις διενεμήθησαν. Η κυρία Λαβίν. Ε, ε, Ευχαριστώ. Στα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών δεν συμφωνούμε. Όταν αποφασίσατε να διαγράψετε τον ε, Αποφασίστε να διαγράψετε τον προσκεκλημένο που είχαμε καλέσει εμείς για μια επόμενη συνεδρίαση και νομίζω ότι ε, έγινε κάποια παρεξήγηση. Εγώ είχα πει όχι, αλλά από ό,τι φαίνεται φάνηκε σαν να είπα ναι. Ε, εμείς υποβάλαμε την πρόσκλησή μας πολύ πριν από την προθεσμία Είχαμε μία πρόταση που ήρθε από τους ε, σοσιαλιστές, την τελευταία στιγμή μάλιστα. Ε, τον, η δική του πρόταση έγινε δεκτή, η δική μας δεν έγινε. Και θέλουμε παρακαλώ τα μέλη να σκεφτούν ε, τι γίνονται αυτέ οι ακροασει. Ο δικός μας προσκεκλημένο, ε, τελευταία στιγμή του το κυρώσαμε και που του είχαμε πει θα έρθει, μετά βλέπαμε δεν θα έρθει. αν μπορούσε να έρθει στις 16 Μαρτίου για να μας μιλήσει για ένα, προ, για ένα πείραμα που έγινε στο, Σκάτ, στο Κάτεγκατ το 2007, θα ήταν ε, καλό. Ούτως ή άλλως εμείς επανερχόμαστε στα ίδια θέματα, διαχείριση των θαλασσών, σάιτης κτλ. Οπότε καλό θα ήταν αν μπορούσαμε στις 16 Μαρτίου να τον έχουμε εδώ κοντά μας αλλά από ό,τι φαίνεται μας βγάλατε τελείως από το πρόγραμμα. Οπότε εμείς δεν θα δεν θα εκπροσωπούμεθα καθόλου σε αυτή την ακρόαση και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Αν η Επιτροπή θέλει όντω να συνεχίσει σε αυτή την άγουσα, πραγματικά εκπλήσωμαι. Και προσωπικά ε, αισθάνομαι θυμό για το ότι πρέπει να τηλεφωνήσω στον προσκεκλημένο και να του πω ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί έγινε παρεξήγηση. Κυρία Λεβίν, δεν, δεν έχω να σας πω κάτι. Αν έγινε παρεξήγηση λυπούμε. Ελήθη όμως η απόφαση και οι υπόλοιποι συμφώνησαν. Ε, αν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε για την απόφαση του πρωινού. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε, δεν δέχεστε αυτό που αποφασίστηκε το πρωί. Ναι, αλλά έγινε μεγάλη συζήτηση σήμερα το πρωί γι' αυτό, κύριο Στίβενσον. Δεν είμαι συντονιστής εγώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα οι συντονιστές έλαβαν την απόφαση εκεί, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς τη συζήτηση. Τώρα, αλλάζουμε τη διαδικασία και οι αποφάσεις δηλαδή των ε, συντονιστών ε, γίνονται αντικείμενο πλήρους συζήτηση στην Επιτροπή. Αν είναι έτσι, γιατί να κάνουμε τη συζήτηση των συντονιστών. Γι' αυτό είπα και εγώ κυρία Λεβίν, ότι όντως έχετε, έχετε κάθε δικαίωμα να υπάρξει ψηφοφορία ε, για την απόφαση αυτή της, ε, των συντονιστών. Αν έχει κάποιος κάποιο επίση ε, πρόβλημα με την πρωινή απόφαση, ας το πει. Λυπούμε πραγματικά που υπήρξε αυτή η παρεξήγηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα να επανέλθουμε. Οπότε να θεωρήσω ότι δεν έχουν υπόλοιπη πρόβλημα, οπότε επιβεβαιώνεται η απόφαση. Ωραία. Άρα η επόμενη συνεδρίαση Βρυξέλλες 15 Μαρτίου και 16 Μαρτίου. Στις συνήθεις ώρες σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος ευχαριστεί και τους δερμηνείς και εμείς καλό σας βράδυ.